Uh, Καλησπέρα. Σημείο 1 της ημερήσιας διάταξης. Ας αλλάξουμε την ημερήσια διάταξη στο σημείο 15. Το 15 το βγάλαμε. Διότι όσον αφορά το μηχανισμό αναστολής και την ψηφοφορία έγινε την περασμένη πέμπτη το σημείο 16 όσον αφορά την σχεδίου εκθέσεως για την καταπολέμηση διαφθοράς και συνέχεια στο ψήφισμα της Ειδικής Επιτροπής ΚΡΙΜ ανεβλήθησαν, ανεβλήθη αυτό. Δύο αλλαγέ λοιπόν, μείον τη 15 και τη 16. Στο σημείο 2, ανακοινώσεις του Προέδρου, δεν έχουμε γοδελικά και ακροατικά δυστυχώς το σήμερα το αύριο. Σημείο 3, έγκριση ημερήσιας διάταξης, με πρακτικά της 1ης Φεβρουαρίου, 21ης-22ης Δεκεμβρίου, 30ης Νοεμβρίου, 1ης Δεκεμβρίου, 12-13 Οκτωβρίου, 15 και 16 Ιουλίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, τα πρακτικά θεωρούνται ως εγκεκριμένα. Πάμε στο σημείο 4. Το πρώτο ουσιαστικό σημείο μας, προστασία της ψηφιακής ιδιωτικότητας ασφαλίζοντας μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ψηφιακή αυτονομία. Θα γίνει ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Γκυγιόμ Πουπάρ, Γενικό Διευθυντή του Γαλλικού Οργανισμού Ασφαλείας των Συστημάτων Πληροφοριών. Θα θυμόσαστε σαν συνέχεια της εκθέσεως για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των υπηκών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στη Λίμπε τον περασμένο Δεκέμβριο διοργανώσαμε μια διάσκεψη υψηλού επίπεδου για την προστασία της ιδιωτικότητας του διαδίκτυου, αυξάνοντας την ασφάλεια του διαδικτύου και τι δυνατότητε που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα διεξήχθη συνεδρίαση μαζί με την Ήτρε, την Ίμκο και τη ΣΤΟΑ. Όπως θα θυμόσαστε, ήταν λεπτομερέστατη η συζήτηση και η διάσκεψη και χρειάστηκε πολύ μενό σχεδιασμό. Ήταν διαδραστική διάσκεψη. 80 εμπειρογνώμονε παγκοσμίου φήμη συμμετείχαν. Βασικέ συστάσει δόθηκαν. Μία από αυτέ ήταν να αναπτύξουμε ισχυρότερο σύστημα, πιο αυτόνομο σύστημα όσον αφορά την πληροφορική στην Ευρώπη το ανέφερα αυτό και το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για την παρακολούθηση του 2014, για τη μαζική παρακολούθηση. Λοιπόν, για να τηρηθεί η όλη ορμή των προσπάθειων και των εξελίξεων, χαίρομαι που έχω σαν φιλοξενούμενο τον κύριο Πουπάρ, που όπως σας είπα είναι ο Γενικός Διευθυντής του Γαλλικού Οργανισμού Ασφαλείας των Σημάτων Πληροφοριών. Άνση. Και προασπίζεται την ε, ευρωπαϊκή αυτονομία στον τομέα και την κυριαρχία. Κύριε Πουπάρ, έχετε το λόγο και είστε ευπρόσδεκτος. Σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για την ασφάλεια την ψηφιακή, κάτι που μας απασχολεί στον οργανισμό από τον οποίο προέρχομαι. Σήμερα θέλω να μιλήσω για την ευρωπαϊκή προσέγγιση, για φιλόδοξους στόχους και να σας υποβάλω και κάποιες ιδέες. Καταρχήν θα επανέλθω στο θέμα της απειλής, έτσι όπως την ε, αντιλαμβανόμαστε στην υπηρεσία την οποία διευθύνω. Βλέπουμε πολλές απειλές, επιθέσεις οι οποίες πολλές φορές μάλιστα δεν ε, δημοσιοποιούνται με σκοπό να προστατεύσουμε τα θύματα αυτών των επιθέσεων. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι με διακατέχει μια σημαντική ανησυχία, διότι βλέπουμε αυτές οι απειλές, αυτές οι επιθέσεις να αυξάνονται, αυτοί οι οποίοι επιτίθενται βελτιώνουν τις τεχνικές τους επιδόσεις, αλλά και αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αυξάνονται αυτές οι επιθέσεις και σε αριθμό αλλά και σε ποιότητα και γίνονται όλο και πιο ε, πολύμορφες. Μιλάμε για την ε, επιθετικότητα στον κυβερνοχώρο, για την εγκληματικότητα με εκλοπές, με επιθέσεις τύπου crypto lockers, οι οποίοι δεν θέλουν απλώς να καταστρέψουν ε, τα δεδομένα με τους παραδοσιακούς ιούς, αλλά με την ψηφιοποίηση της ε, πληροφορίας και κατόπιν ζητούν από τα θύματα έναντι λίτρων τα οποία μάλιστα του ζητούν να πληρώσουν με ένα νόμισμα τύπου bitcoin και με κάποιες χιλιάδες ευρώ, αν θέλετε, συνήθως αυτοί οι εγκληματίες σας επιτρέπουν να ξαναέχετε πρόσβαση στα δικά σας δεδομένα. Πρόκειται λοιπόν για διάφορες επιθέσεις. Κάποιοι μάλιστα μέχρι τώρα έχουν ε, δεχθεί αυτές τις ε, συναλλαγές, έχουν πληρώσει, χωρίς όμως καμία εγγύηση αν θέλετε για να μπορέσουν να ξανέχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους. Πρόκειται για διεθνείς σπήρες, διεθνείς εγκληματίες και κανείς δεν ξέρει τι κάνουν με αυτά τα χρήματα. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένος ότι αυτά τα χρήματα επανεπενδύονται για την ε, περαιτέρω ανάπτυξη τέτοιων πρακτικών παράνομων και εγκληματικών. Το δεύτερο πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι κάτι που παρατηρείται όλο και πιο συχνά. Είναι η δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων πληροφοριών. Δηλαδή άνθρωποι που προσπαθούν να διεισδύσουν στα ιδιωτικά και τα δημόσια δίκτυα σε μεγάλες επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις με πολύ πολύτιμες πληροφορίες, τη διοίκηση και προσπαθούν να υποκλέψουν δεδομένα εμπορικού χαρακτήρα, τεχνικού χαρακτήρα. Οτιδήποτε λοιπόν μπορεί να αποτελέσει τον πλούτο μιας επιχείρησης. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα είναι ένα συνήθες φαινόμενο, το οποίο βεβαίως πολλές φορές δεν έχει αναγνωριστεί η σωστή του αξία ένας ε, ο οποίος έχει πρόσβαση ή παράνομα σε ένα τέτοιο δίκτυο, καταρχήν θέλει να μην τον αντιληφθούν, να μην εντοπιστεί. Εάν λοιπόν δεν εντοπιστεί ο συγκεκριμένος ε, εγκληματίας, Μπορεί μια επιχείρηση να μην αντιληφθεί καθόλου ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ στη δική μου υπηρεσία εντοπίσαμε περίπου 20 τέτοιες επιθέσεις πέρσι, δηλαδή κατά σημαντικών φορέων της γαλλικής οικονομίας, από τους οποίους υπεξαιρέθηκαν πολύ σημαντικά δεδομένα, πληροφορίες και Πραγματικά σας λέω για άλλη μια φορά ότι ανησυχώ ιδιαίτερα. Εντοπίσαμε, όπως σας είπα, περίπου 20 τέτοιες περιπτώσεις. Δεν μπορώ όμως σε καμία περίπτωση να σας δώσω τον πραγματικό αριθμό αυτών των επιθέσεων, καθότι τις περισσότερες δεν τις έχουμε εντοπίσει, άρα δεν ξέρουμε πόσες είναι. Επίσης, ποιος ε, ε, είναι πίσω από αυτές τις ε, επιθέσεις. Ειλικρινά δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν πρόκειται για κράτη, αν πρόκειται για φορείς που βρίσκονται στον βορρά, στον νότο, στην Ανατολή, στη Δύση, αν πρόκειται για ομάδες τύπου μαφίας, αν πρόκειται για ανταγωνιστές και στις περισσότερες από τις έρευνες που κάνουμε από κοινού με τις υπηρεσίες πληροφοριών και την αστυνομία, διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές πρόκειται για οργανισμούς που καμιά φορά εργάζονται για κάποιο κρατικό φορέα, όμως μπορεί κάλλιστα να εργαστούν και μόνοι τους ή για λογαριασμό κάποιας εγκληματικής οργάνωσης. Τρίτη απειλή είναι αυτή του σαμποτάζ. Και σήμερα φοβόμαστε ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να υποκλέψει πληροφορίες χωρίς να αλλοιώσει καθόλου τα δίκτυα θα μπορούσε ενδεχομένως με τον ίδιο τρόπο να πλήξει τη λειτουργία, την εύρυθμη λειτουργία αυτών των δικτύων, να παρεμποδίσει τις δραστηριότητες και ενδεχομένως να διεισδύσει σε δίκτυα χωρίς ε, συγκεκριμένα δεδομένα, αλλά να πλήξει, παραδείγματος χάρη, πολύ σημαντικές υποδομές, όπως τα δίκτυα μεταφορών, δηληστήρια, βιομηχανίες. Καταλαβαίνετε, παραδείγματο χάρη, ότι η καλή λειτουργία ενός δηληστηρίου που σήμερα λειτουργεί με ψηφιακό τρόπο και ελέγχεται με ψηφιακό τρόπο, είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι επιτίθενται μπορεί να έχουν ε, πολιτικούς ή οικονομικούς ε, σκοπούς, μπορεί να προκαλέσουν ε, καταστροφή. Καταλαβαίνετε τι μπορεί να προκαλέσει κανείς αν ελέγξει, παραδείγματος χάρη, τις ε, σιδηροδρομικές γραμμές, τα δίκτυα ενός ε, κράτους. Σήμερα έχουμε, αν θέλετε, λίγες τέτοιες επιθέσεις και αυτό βεβαίως δεν οφείλεται στην ε, σημαντική τεχνολογία που διαθέτουμε για να τις αποτρέψουμε, αλλά ενδεχομένως στην έλλειψη τέτοιων επιθέσεων. Όπως ξέρετε υπήρξε η επίθεση κατά του καναλιού TV5 και μάλιστα ξέρουμε σήμερα ότι έγινε η προσπάθεια ότι ο επιτιθέμενος έφτασε μάλιστα μέχρι την τελευταία φάση της επίθεσης ήταν έτοιμος να καταστρέψει όλο το δίκτυο. Σήμερα δεν ξέρουμε ακόμα ποιες ήταν οι συγκεκριμένες βλέψεις αυτού του εγκληματία και ξέρουμε ότι βεβαίως τέτοιου είδους επιθέσεις μπορεί να έχουν και πολύ πιο ε, συγκεκριμένα αποτελέσματα και πολύ πιο ε, σοβαρά αποτελέσματα, ακόμα και θύματα, ανθρώπινες ζωές ε, και τραυματίες. Οι κοινωνίες μας λοιπόν οφείλουν σήμερα να αντιδράσουν. Είναι καθήκον των δημοκρατικών μας ε, πολιτευμάτων να κινητοποιήσουν όλα τα συστήματα προστασίας και ασφαλείας. Μπορούμε να το κάνουμε, έχουμε την απαραίτητη τεχνολογία, είναι θέμα ψηφιακής ασφάλειας και σήμερα γνωρίζουμε ότι η ψηφιακή ασφάλεια δεν είναι αποκλειστικά θέμα κάποιων ειδικών εμπειρογνωμόνων, αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μας απασχολήσει όλους. Ο καθένας στο επίπεδό του θα πρέπει να αναρωτηθεί πώς μπορούμε να προστατευτούμε με συλλογικό τρόπο έναντι αυτών των ε, κυβερνοεπιθέσεων. Στη Γαλλία δημιουργήσαμε αυτή την υπηρεσία την οποία εγώ διευθύνω. Η ΑΝΣΥ ιδρύθηκε το 2009. Ήμασταν 100 άτομα, σήμερα είμαστε 500 στην ΑΝΣΥ. μας στηρίζει το γαλλικό κράτος. Οι απειλές και οι επιθέσεις στο κυβερνοχώρο λαμβάνονται πολύ σοβαρά από την γαλλική δημοκρατία και βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη μας όλες αυτές τις επιθέσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας. Και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι υπηρεσίες πληροφοριών να ε, αναλάβουν το σύνολο αυτής της προστασίας γιατί είναι πιο λογικό και από άποψη τεχνική. Από την άλλη βεβαίως υπάρχουν αντικρώμενα συμφέροντα και σε κάθε περίπτωση εγώ προσέχω ιδιαίτερα όλες τις πληροφορίες που φτάνουν ως εμένα από τις υπηρεσίες πληροφοριών. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι επιθέσεις, αν θέλετε, προετοιμάζονται ή ενδεχομένως θα συμβούν. Όμως, η αρχική μου αποστολή είναι η προστασία των ε, θυμάτων. Από την άλλη, και αυτό ίσως είναι μια γαλλική προσέγγιση, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, έχουμε την ε, βούληση με κανονισμούς και ρυθμίσεις να κερδίσουμε χρόνο και να προλάβουμε αυτούς τους επιτιθέμενους. Σκοπός μας είναι επίσης να προστατεύσουμε τους πιο αδύναμους φορείς. Η ψηφιακή ασφάλεια δεν είναι σήμερα επιλογή, είναι μια υποχρεωτική λύση. Και από το Δεκέμβριο του 2013 με την πρώτη νομοθεσία και την εφαρμογή της η οποία συγκεκριμενοποιεί ε, με τις εφαρμοστικές διατάξεις αυτή την νομοθεσία και με αυτόν τον τρόπο η η υπηρεσία μου, μπόρεσε να προστατεύσει αυτούς τους πιο ευάλωτους ε, φορείς, να εκτιμήσει και να αξιολογήσει σωστά τις απειλές. Μας επέτρεψε επίσης να προετοιμάσουμε από κοινού κανόνες έτσι ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ως προς την προστασία. Αυτά τα κάναμε τα δύο τελευταία χρόνια. Πριν από 15 μέρες βγήκε η τελευταία διάταξη και η λεγόμενη ζωτική σημασίας οργανισμοί και φορείς, τους οποίους καλούμαστε να προστατεύσουμε. Βάσει αυτών των κανόνων θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους και στο σωστό επίπεδο αυτήν την κυβερνό ασφάλεια με θέματα που άπτονται της διακυβέρνησης και αυτό βεβαίως αφορά όλους τους επικεφαλείς και των ιδιωτικών αλλά και των δημόσιων φορέων. Σκοπός μας δεν είναι να προσθέσουμε επιπλέον ρυθμίσεις και κανονισμούς, αλλά να συνειδητοποιήσουν οι ηγεσίε όλων αυτών των οργανισμών την ανάγκη προστασίας με φιλόδοξο τρόπο. Και αυτό σε όλους τους τομείς, και στις μεταφορές και στην ενέργεια και στην, στο θέμα του το χρηματοπιστωτικό τομέα και στα δίκτυα το νερό κτλ. Υπάρχει λοιπόν μια εθνική προσέγγιση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι όλα αυτά τα δίκτυα, όλοι αυτοί οι μεγάλοι φορείς και οργανισμοί δεν σταματάνε στα γαλλικά σύνορα και υπάρχει πολύ σημαντική ε, αλληλεπίδραση. Παράδειγμα, με την ενέργεια, την ε, ηλεκτρική ενέργεια, παράγουμε και διανέμουμε ηλεκτρισμό, αλλά σε κάθε περίπτωση εξαρτόμαστε και από τη δυνατότητα των γειτονικών χωρών να πράξουν το ίδιο. Και σε κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ότι η αδυναμία ή το πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας εταίρος μας θα έχει επιπτώσεις και σε μας. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι περισσότεροι φορείς είναι ήδη ευρωπαϊκοί φορείς, είτε πρόκειται για οργανισμούς ε, που συνεργάζονται Γι' αυτό και χαιρετίζω την οδηγία ΝΙΣ, η οποία αφορά την ασφάλεια των δικτύων και θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και να μην περιοριζόμαστε σε εθνικά μέτρα. Λέγατε, κύριε Πρόεδρε, ε, ότι υπάρχει και η έννοια της αυτονομίας, της στρατηγικής αυτονομίας. Εγώ είμαι υπέρμαχος ε, αυτής της στρατηγικής αυτονομίας. Θα σας εξηγήσω σε λίγο τι ακριβώς σημαίνει. Η στρατηγική αυτονομία, έτσι όπως την αντιλαμβανόμαστε στη Γαλλία, δεν σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε προστατευτικά σύνορα και ότι δεν πρέπει να συνεργαζόμαστε με άλλους ξένους φορείς. Και εδώ αναφέρομαι βεβαίως στις αμερικανικές ε, εταιρικές, ε, σε αμερικανικές εταιρικές σχέσεις που ενδεχομένως μπορούμε να έχουμε. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποιους τομείς, να ελέγχουμε κάποιες τεχνολογίες και να μην περιμένουμε την καινοτομία και τους κανόνες που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρώπης. Αυτή η στρατηγική αυτονομία λοιπόν στηρίζεται κυρίως στην ανάγκη να διασφαλίσουμε εμείς την ψηφιακή μας ασφάλεια. Δεν μπορεί μια χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διασφαλίσει ε, με μία προστασία του κυβερνοχώρου την Ευρώπη ή κάποιες χώρες της Ευρώπης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν έχει νόημα και θα πρέπει η κάθε χώρα να αναλάβει την ασφάλεια του κυβερνοχώρου της και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το θέμα αυτό. Χαιρετίζω την θέσπιση του CERTU γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πληροφορικές απειλές και επιθέσεις όπως και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Λέντιζα, η Ένιζα, η οποία είναι αν θέλετε ο αντίστοιχος φορέας με την δική μας υπηρεσία στη Γαλλία και βεβαίως θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο και σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ο υπολογισμός αυτής της υπηρεσίας σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ανεπαρκής. Πολύ αδύναμος προϋπολογισμός εν ώψη των απειλών που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ο νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής της ε, Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας εξελέγει πρόσφατα, προέρχεται από την ΑΝΣΥ, είναι Γάλλος και η συνεργασία μεταξύ της ΑΝΣΥ και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σίγουρα ε, δεν μπορεί παρά να ενδυναμωθεί από εδώ και πέρα. Πέρα από την προστασία των κρατών των ευρωπαϊκών θεσμών, θα πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα της ε, βιομηχανικής ανεξαρτησίας. Κάτι που δεν σημαίνει ότι κλεινόμαστε στον εαυτό μας και ότι δεν συνεργαζόμαστε με βιομηχανίες εκτός της ε, Ευρώπης. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση όμως στον ψηφιακό τομέα, στον τομέα του κυβερνοχώρου, να αναπτύξουμε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα Έχουμε σημαντικούς φορείς και είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να ελέγξουμε αυτήν την τεχνολογία, την ψηφιακή ασφάλεια. Υπάρχουν τέτοιοι φορείς ήδη στην Ευρώπη, πρέπει να τους στηρίξουμε, πρέπει να τους δώσουμε κίνητρα και ίσως να ξανασκεφτούμε τον ψηφιακό τομέα, πως παραδείγματο χάρη αγοράζουμε προϊόντα στα κράτη-μέλη, στην Ευρώπη ίσως να επιλέξουμε πιο ασφαλή προϊόντα και συστήματα, τεχνολογίες πιο ασφαλείς, τα λεγόμενα ελεύθερα λογισμικά, τα οποία χωρίς να έχουν 100% ασφαλή αποτελέσματα, έχουν πολύ περισσότερη αν θέλετε, ε, προστασία και υψηλό, προσφέρουν υψηλότερη ασφάλεια. Το θέμα επίσης της πιστοποίησης πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα συστήματα που αγοράζουμε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη και οι επιχειρήσεις μας πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη. Αυτό προϋποθέτει πιστοποίηση. Πιστοποίηση προϊόντων, συστημάτων, ευρωπαϊκών και μη ευρωπαϊκών και χρειάζονται ασφαλείς έλεγχη για όλα αυτά τα συστήματα εμπιστοσύνης πρέπει να μπορούμε να διεισδύσουμε και να δούμε τι ακριβώς ε, περιεχόμενο έχουν για να μπορούμε να τα πιστοποιήσουμε. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί την προηγούμενη εβδομάδα υπεγράφει μια εταιρική σχέση δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εμείς Βεβαίως ε, ανήκουμε σε αυτήν την ε, εταιρική σχέση. Υπάρχουν κονδύλια που θα διατεθούν για την έρευνα και την ανάπτυξη και αυτό επίσης το θεωρώ εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να σας παρουσιάσω είναι η ανησυχία μου, ο φόβος μου στο μέλλον να μην μπορούμε πλέον να ρυθμίσουμε τον τομέα του κυβερνοχώρου και αυτό στα πλαίσια των εμπορικών ε, διαπραγματεύσεων όπως το ΤΙΖΑ, το ΤΙΤΙΠ γιατί αυτά που αναλαμβάνουμε για το θέμα της ασφάλειας μπορεί να θεωρηθούν εμπορικά εμπόδια. Σε καμία περίπτωση δεν είναι. Σκοπός μου είναι η ασφάλεια και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπορούμε στην Ευρώπη να συνεχίζουμε να νομοθετούμε, να θεσπίζουμε μέτρα και κανόνες γιατί αυτό είναι απαραίτητο για την ασφάλειά μας. Μπορεί κάποιοι να το θεωρήσουν εμπόδιο, ε, πραγματικά όμως πρέπει να συνεχίσουμε να μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά την ψηφιοποίηση θα πρέπει να μπορούμε να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτήν την τεχνολογία, την τεχνολογία της κρυπτοποίησης με σκοπό να κωδικοποιήσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε ε, συγκεκριμένα δεδομένα τα οποία θα πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικά, να προστατεύονται για να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση εγκληματικές οργανώσεις, τρομοκράτες κτλ. Όσον αφορά τις επικοινωνίες, Βεβαίως και θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων μας και της ασφάλειας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουπά. Ε, θα δώσουμε το λόγο στους ομιλητές για κάποιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπόνι για αυτή την ε, πλήρη παρουσίαση. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυξάνεται ο ρόλος του κυβερνοεγκλήματος δυστυχώς και πρέπει να υπάρχουν ε, καταλληλότερες απαντήσεις. Και συμφωνώ τα μαζί σας όταν ε, μας λέτε ότι οι λύσεις της ψηφιακής ασφάλειας θα πρέπει να είναι υποχρεωτικές για όλους τους ε, εταίρους, για όλους τους τομείς, ιδίως όταν αναφερόμαστε σε κρίσιμες υποδομές, αλλά όχι μόνον για αυτές. Τώρα βρισκόμαστε στο διάστημα της εφαρμογής της ε, οδηγίες ε, για τα πληροφορίες των δικτύων και την ασφάλεια. Η επιτυχία της εφαρμογής αυτής της οδηγίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον υπάρχει διάθεση για συνεργασία, ε, πραγματική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Τι άποψη έχετε εσείς, διότι στη διάρκεια της ε, κατάρτισης της οδηγίας ε, νης συζητήσαμε τι μπορεί να γίνουν και κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν. Υπάρχουν κάποια προσκόμματα και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία. Θεωρώ ότι στο μέλλον και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε τώρα αυτό, ότι μπορούμε να συζητήσουμε για την ασφάλεια ως αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά όταν συζητούμε την ψηφιακή ασφάλεια που είναι εκφύσεως ε, ε, διεθνής, θα πρέπει να είναι ε, θέμα ευρωπαϊκής αρμοδιότητας και να μην είναι μόνο στα χέρια των κρατών μελών. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Και η δεύτερη ερώτησή μου αφορά το κατά πόσον αυτή η πολιτική για την κυβερνοασφάλεια θα είναι πολύ πιο ε, ρεαλιστική για διάφορους λόγους. Μπορεί να είναι ισχυρότερη η κυβερνοασφάλεια μέσω άλλης συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών, θεσμικών οργάνων και κρατών μελών, μέσω κατάλληλης νομοθεσίας, μέσω τεχνολογίας, ε, security by design όπως το λέμε, Αναφερθήκατε στην κρυπτογράφηση και νομίζω ότι θα πρέπει να τη συζητήσουμε την κρυπτογράφηση, αλλά πρέπει να συζητήσουμε και τα θεμελιώδη δικαιώματά μας ε, στην προστασία της ιδιωτικής μας ζωής. Η κρυπτογράφηση λοιπόν για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Και κάτι τελευταίο θα πρέπει να αναπτύξουμε την κατανόηση της κυβερνοασφάλειας μέσω προώθησης όλων αυτών των συστημάτων. Επομένως, η σχετική οδηγία θα μας παρέχει και κάποια εργαλεία για την προώθηση όλων αυτών των θεμάτων, πώς μπορούν ε, να έχουμε και συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλες αυτές τις δραστηριότητε. Ευχαριστώ, κυρία Σύπρου. Ευχαριστώ. Εγώ παρακολούθησα όλες αυτές τις συζητήσεις και στο παρελθόν και σήμερα για την προστασία των δεδομένων. Είπατε ότι θα πρέπει να κερδίσουμε χρόνο και να προτρέξουμε όλων αυτών των εγκληματιών. Δεν είμαι όμως τόσο σίγουρη ότι μόνο αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί σήμερα υπάρχουν ε, έργα βιβλία που αναφέρουν όλη αυτή την κούρσα, την ε, τεχνολογική. Το θέμα της ε, προστασίας ε, των δεδομένων, της κωδικοποίησης, πρέπει ή δεν πρέπει. Γιατί από τη μία είναι η προστασία για να μην χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και από την άλλη βεβαίως υπάρχει ο οικονομικός ανταγωνισμός και τα εμπόδια στην οικονομία. Το θέμα είναι όμως ότι αν θέλουμε τέτοιου είδους προστασία δεν θα πρέπει να αφήσουμε ούτε μαχαίρια κουζίνας, γιατί και αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εγκληματίες και από τρομοκράτες. Μπορείτε να μας πείτε λοιπόν πού ξεκινάει το ευρωπαϊκό επίπεδο σε όλα αυτά. Γιατί εδώ, όπως είπατε, είναι και θέμα χρηματοδότηση. Είναι θέμα αν αυτά τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για να διατεθούν για αυτό τον τομέα. Σήμερα πείτε μου συγκεκριμένα τι γίνεται σε εθνικό, σε περιφερειακό επίπεδο, γιατί κάπου πρέπει να κλείσουμε αυτά τα δίκτυα, να κλείσουμε αυτές τις ροές, έτσι ώστε να μην περνάει τίποτα σε περιοχές, σε κράτη. Αναρωτιέμαι λοιπόν πού είναι οι επενδύσεις, πού είναι οι επενδύσεις, πού είναι τα κίνητρα για να προστατευτεί ο ίδιος ο ιδιωτικός τομέας, ο, οι ίδιες οι επιχειρήσεις, να μην υπάρχουν επιθέσεις προς τις ε, επιχειρήσεις. Σήμερα ξέρουμε ότι πολλοί συγκεκριμένες επιχειρήσεις κάνουν πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα κάνουν. Χρησιμοποιούν ρομπότ, τεχνολογίες στην βιομηχανία παραδείγματος χάρη. Μπορείτε να μου πείτε τι θα γινόταν αν ένα τέτοιο σύστημα ρομποτικό, τεχνολογικό που έχουμε στα αυτοκίνητά μας ε, ήταν ε, κάτι το οποίο θα χειριζόταν εγκληματικές οργανώσεις, καταλαβαίνετε τα αποτελέσματα και για τις μεταφορές και για άλλους τομείς όπως τα δίκτυα ενέργειας. Αυτό λοιπόν που ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει σήμερα είναι να δούμε και όσον αφορά την προστασία ε, παραδείγματος χάρη ενός καναλιού ή ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Γιατί είναι αντικείμενο επίθεσης. Γιατί η, η προπαγάνδα κάποιων φορέων και κάποιων εγκληματιών δεν φτάνει να περνάει από τα κοινωνικά δίκτυα, από το διαδίκτυο. Γιατί πρέπει να περάσει και από τα τηλεοπτικά κανάλια ή τους ροδιοφωνικούς σταθμούς. Εγώ πάντως επιμένω ότι για να αυξηθεί η προστασία και η ασφάλεια χρειάζονται περισσότερα κονδύλια, περισσότερη χρηματοδότηση. Είναι σίγουρα θέμα ευαισθητοποίησης, θα πρέπει και οι ίδιες επιχειρήσεις ή διάφοροι βιομηχανικοί τομείς να προστατεύσουν τον εαυτό τους, αλλά την ίδια ώρα να συνειδητοποιήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι πολλά μπορούμε να κάνουμε και κάθε νέα τεχνολογία εμπεριέχει νέους κινδύνους με τους οποίους θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε. Κυρία Ιντβελτ, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και που πάγια την παρουσίασή σας. Τι να σας πω όμως, με κάπως με αυτά που άκουσα, που είπατε. Στο τέλος της παρέμβασής σας είπατε ο ίδιος ότι δεν θέλετε να διαδώσετε ένα αποστατευτισμό Αλλά νομίζω ότι σε όλη την παρέμβαση αυτήν την τύπωση σχημάτισα. Δεν είναι θέμα για, αυτό, για αυτονομία, δεν αφορά την αυτονομία και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό που προτείνεται είναι ένα τείχος γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η διάδραση με άλλα μέρη του κόσμου θα γίνει δυσχερέστερη. Εγώ από τα πράγματα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ισχυροποιηθεί η ίδια. Ο νέος Steve Jobs θα πρέπει να είναι Ευρωπαίος. Πώς θα το πετύχουμε αυτό. Εξαλείφοντας τους φραγμούς στην εσωτερική αγορά. Κάτι που δεν υποστηρίζει πάντα η γαλλική κυβέρνηση. Το άλλο στοιχείο, έχουμε πάρα πολλούς κανονισμούς, κανέναν, κανένας δεν τον εφαρμόζει. Θα μιλήσαμε για την προστασία της ιδιωτικότητας. Εγώ προσωπικά είμαι πεπισμένη ότι δεν, είναι, δεν αντέχει τις δοκιμασίες περί νομιμότητας και καθαταρεύσει ενώπιν των δικαστηρίων. Δεν μπορούμε να βασιστούμε στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκλειστικά να επιβάλλουν και να στηρίξουν τους νόμους μας. Και αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό, τότε μπορούμε εσαΐ. Μέχρι τελικής πτώσεως νομοθετούμε και δεν θα είμαστε ασφαλέστεροι παρουσιάζεται το TTIP σαν ένα τέρα, σαν μια απειλή που στρέφεται κατά της ασφαλείας των ευρωπαϊκών συστημάτων. Εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη απειλή είναι η κακή εφαρμογή των νόμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η κυβέρνησή σας ενέκρινε την συμφωνία ομπρέλα που υπονομεύει την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια αυτών. Στηρίζει επίσης και απαγόρευση κρυπτογράφησης και ανοιχτών θυρών πρόσβαση στο λογισμικό. Και έχει πάρα πολύ, έχει θεσπίσει νομοθεσία που παραβιάζει την ιδιωτικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σωστά περιγράφεται βέβαια τους κινδύνους και το ότι όλοι πρέπει να τους γνωρίζουμε. Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι. αν δείτε ένα μεγάλο χακάρισμα που έγινε πριν από δύο χρόνια. Δηλαδή, οι μυστικές υπηρεσίες Βρετανίας παραβίασαν το σύστημα της Belgacom και μετά από τρία χρόνια σιωπής οι βελικές δικαστικές αρχές συνεπέραναν ότι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι έγινε παραβίαση. Άρα ε, ακυρώθηκε η όλη δικαστική προσπάθεια. Εντάξει, καλό να λέτε ότι πρέπει να είμαστε εξάρτητοι, αλλά και τον με τείχο γύρω από την Ευρώπη δεν με καθησυχάζει. Λοιπόν, αντί να μιλάμε για προστατευτικά μέτρα, ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα έλεγα ότι τι σημαίνει να αυξήσουμε τη δυνατότητα που θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να αμυνθεί, να εξαρτώνται λιγότερο οι εταιρείε μας από τις εταιρείε τρίτων χωρών και θα πρέπει να επιβάλλουμε τους θεσπιστέντες κανόνες. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Δεν θέλουμε να απομονωθούμε. Δεν θέλουμε συνεχώς να τελούμε να μείνει, αλλά να επιθέσει επίσης. Ευχαριστώ κυρία Λόρεστον. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Σημαντικότατο θέμα. Όλοι το κατανοούμε. Πρέπει να το συζητήσουμε σοβαρά, ξεκινώντας από τις βάσεις. Τι εννοούμε με κυβερνοασφάλεια με τη λέξη αυτή, μέχρι πού το φτάνουμε και πώς θα κάνουμε σωστή διαφοροποίηση των διαφόρων στοιχείων της ασφαλείας και των στοιχείων που άπτονται της εθνικής ασφαλείας. Εγώ είμαι στον Ι. Έχουμε κέντρο κυβερνοασφαλείας για το ΝΑΤΟ. Λειτουργεί για την προστασία του ΝΑΤΟ προβληματίστηκα. Ίσως να μην κατάλαβα καλά, αλλά προβληματίστηκα με αυτό που άκουσα. Είπατε ότι μάλλον πρέπει να ψώσουμε τείχος μεταξύ κυβερνοασφαλείας με τους συμμάχους μας σε παγκόσμιο επίπεδο, με το ΝΑΤΟ, να έχουμε αυτό από τη μία και να έχουμε ευρωπαϊκή κυβερνοασφάλεια που θα είναι διαφοροποιημένη. Δύο συστήματα δηλαδή. Ένα για όλους, συμμάχους στο ΝΑΤΟ και ένα για την Ευρώπη. Αυτό με προβληματίζει. Μπορείτε να το διευκρινίσετε, Τώρα απ' την άλλη, βλέποντας την καθημερινή ασφάλεια. Δεν νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μόνο με αυστηρή νομοθεσία και με εθνικούς ή διεθνείς κανόνες και μόνο. Βλέποντας τα περιστατικά. Στην Εστονία δεχτήκαμε επιθέσεις, έχουμε εμπειρία κυβέρνων επιθέσεων από τους άλλους, από τις άλλες τρίτες χώρες, κάποιες άλλες τρίτες χώρες. Και τι είδαμε ότι πολλά γίνονται σε ιδιωτικό επίπεδο. Οι hackers χρησιμοποίησαν τα διάφορα δίκτυα. Υπήρχε και άμυνα. Σε επίπεδο πολιτών, όχι κράτους. Σε επίπεδο κοινοτήτων του κυβερνοχώρου και αυτό ήταν πιο αποτελεσματικό από ένα το εθνικό σύστημα στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη. Πώς μπορούμε να κάνουμε να συμμετάσχουν οι πολίτες, αποκτώντας δεξιότητες, γνώσεις. Υπάρχει μεγάλη διαφορά από χώρα σε χώρα, μεγάλη διαφορά. Και πρέπει να επαγρυπνούμε, να καταλάβουμε ότι το κλειδί στην ασφάλεια είναι στον υπολογιστή του καθενός και έχει σε κάποιο κυβερνητικό κτίριο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Έχω μία ερώτηση, εδώ πίσω είμαι εγώ. Για τα μέτρα ασφαλείας στην πληροφορική. Και βάσει τον όσων είπε ο κύριος Μπόνι. Έχουμε την οδηγία για την ασφάλεια των δικτύων που αφορά τα διάφορες, διάφορες κρίσιμες υποδομές κατά πόσο πρέπει να έχουμε γενικές προδιαγραφές για τα συστήματα πληροφορικής. Κανόνες περί ευθυνών των παραγωγών των τεχνολογιών. Διότι θα είναι και πιο δύσκολο να εξασφαλίζεται η ασφάλεια από έναν. Και θα πρέπει να προβλέπονται και κυρώσεις για κάποιες ευθύνες όταν υπάρχουν αποδεδειγμένες ζημίες και βλάβες. Δύσκολο όμως να αποδειχθούν οι βλάβες που προκύπτουν από κάποια κενά. Τα κενά δημιουργούν προβλήματα. Άρα πρέπει να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να καλύπτει τα κενά. Ευχαριστώ πολύ Γιάν Κάποιος άλλος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου. Θεωρώ ότι ήταν πολύ καλή η συνεδρία σε αυτή. Θέλαμε να δώσουμε έναυσμα για αυτά τα θέματα μετά από τις διάφορες συζητήσεις που είχαμε και την έκθεση για τη μαζική παρακολούθηση και τις ακροάσεις που κάναμε. Και θα ήθελα να κάνω και μια σύντομη ερώτηση. Μπορεί να μην έχετε χρόνο βέβαια να απαντήσετε σε όλες. Μετά από την ερώτηση για την οδηγία νης, ε, την οποία αναφέρατε εσείς πρώτος, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό ερώτημα που τέθηκε στην ε, διάσκεψη ψηλού επίπεδου και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν σαφές. Μπορεί να έγινε και σκεμμένα αυτό γιατί είναι δύσκολο το ερώτημα. Προτείνεται ότι επειδή δεν ε, έχουμε φραγμούς, δεν προσπαθούμε να έχουμε νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως δεν έχουμε και σχετική νομολογία για τα θέματα πληροφορικής και τελικά ε, δεν μπορούμε να έχουμε νέες δυνατότητες και άρα κατά κάποιο τρόπο δημιουργούμε φραγμεούς γιατί δημιουργούμε μια νέα ευρωπαϊκή δομή δεν θα έχουμε άμυνα, αλλά θα έχουμε νέε δυνατότητε και θα έχουμε ισχύ από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα γίνει μέσω νομοθεσία και αναφερθήκατε κι εσεί στην νομοθεσία και ε, φαίνεται ότι αυτή είναι η σωστή άκουσα. Θα ήθελα να ξέρω εσεί τι βλέπετε ότι πρέπει να κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε του πολίτε δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε εσκεμμένα ένα αντίβαρο προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτό προτείνετε εσείς, για να καταλάβουμε λίγο προς τα πού οδεύουμε. Διότι όλοι ξέρουμε ότι η νέα οδηγία είναι καλή και όλοι αντιλαμβανόμαστε τι πρέπει να κάνουμε με αυτή την νομοθεσία, αλλά εσείς προς ποια κατεύθυνση θεωρείτε ότι θα πρέπει να ε, κινηθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αν καταλαβαίνω εγώ καλά, δεν θα δημιουργήσουμε εμείς ε, φράγματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να προστατευτούμε με διαφόρους τρόπους. Θα ήθελα να ξέρω τι έχετε να μας πείτε εσείς. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω μέσα στο χρόνο που διαθέτω, αν και δεν έχω πολύ χρόνο. Η οδηγία νης την οποία αναφέρατε πολλές φορές και εσείς, ε, την ανέφερα και εγώ, είναι σημαντική για μας γιατί ουσιαστικά εκπέμπει ένα μήνυμα προς τα κράτη-μέλη, κυρίως αυτά που ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει το τι πρέπει να γίνει για θέματα ασφάλειας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό η συνεργασία σε δίκτυο. Όπως ε, πολύ σωστά είπατε, οι κρίσιμες υποδομές ξεπερνούν τα σύνορα ενός κράτους μέλους. Πρόκειται για θέματα που είναι ζωτικής σημασίας, που αφορούν πολύ συχνά θέματα εθνικής κυριαρχίας και όταν εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε κάποια θύματα επιθέσεων, διαπιστώνουμε ότι πρόκειται καθαρά για θέματα που άπτονται της ασφάλειας των κρατών μελών. Αυτοί που επιτίθενται βεβαίως δεν κάνουν τέτοιου είδους διακρίσεις. Μπορούν να επιτεθούν κατά μιας επιχείρησης στον αμυντικό τομέα και κατόπιν να περάσουν σε μια επιχείρηση ενός άλλου τομέα, χωρίς να κάνουν ε, τέτοιου είδους διακρίσεις και κατηγοριοποιήσεις θυμάτων. Η έννοια του δικτύου σαν πρώτο μοντέλο συνεργασίας είναι για μένα πολύ σημαντικό. Οι μέχρι τώρα επαφές που είχα με φορείς άλλους κρατών μελών, άλλων κρατών μελών, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πραγματικές επιθέσεις, για πραγματικά θύματα, δεν είναι εύκολο να γίνουν οι συζητήσεις σε άλλο επίπεδο από το διμερές. οι πιο πολλοί δεν θέλουν να ενημερώσουν όλους τους εταίρους όταν έχουν υποστεί τέτοιες επιθέσεις. Ξεκινάμε λοιπόν με το μοντέλο αυτό του δικτύου σε διμερές επίπεδο. Αν προσπαθήσουμε όλα τα κράτη-μέλη να συζητήσουν για αυτού του είδους τα εμπιστευτικά θέματα, πολύ φοβάμαι ότι θα παραμείνουμε σε ένα πολύ αναποτελεσματικό και ε, επιφανειακό επίπεδο. Μου κάνατε επίσης την ερώτηση για τις ε, συγκεκριμένες πολιτικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Σήμερα ξέρουμε να προστατευτούμε, ξέρουμε να αναπτύξουμε συστήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, να προστατεύσουμε τις πληροφορίες, τα δεδομένα να προετοιμάσουμε συστήματα που θα αποτρέψουν τέτοιου είδους επιθέσεις με τη χρήση τεχνολογίας κρυπτογράφησης. Μπορούμε επίσης να εντοπίσουμε τις επιθέσεις, αν και ακόμα και σήμερα πολύ λίγοι ανοιχνεύουν αυτές τις επιθέσεις με τρόπο αποτελεσματικό. 100% αποτελεσματικότητα δεν υπάρχει σε κανένα σύστημα. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία και η συνεργασία σημαίνει διασύνδεση μεταξύ των δικτύων και σημαίνει ότι πάντα θα υπάρχει δυνατότητα για κάποιον κακόβουλο να διεισδύσει. Από την άλλη υπάρχει όπως είπατε και το θέμα της ευαισθητοποίησης των ε, ανθρώπων. Πρόκειται για πληροφορική, η πληροφορική βεβαίως προϋποθέτει ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται δεδομένα που αφορούν τους πολίτες. Ο καθένας λοιπόν στο επίπεδο του, οι χρήστες στο επίπεδο των χρηστών, οι ηγέτες και οι αρχές στο δικό τους επίπεδο και με την στήριξη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Συστημάτων θα πρέπει να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όλων. Αναφερθήκατε σε πολλές ενδιαφέρουσες περιπτώσεις για τις οποίες θεωρείτε ότι είμαστε καθυστερημένοι. Μιλήσατε για πιθανούς στόχους. Και αυτές οι καθυστερήσεις είπατε οφείλονται και σε σημαντική έλλειψη επενδύσεων από μέρους των κρατών μελών. Κανείς στην Ευρώπη, αλλά και εκτός Ευρώπης, δεν μπορεί να πει ότι είμαι απολύτως προστατευμένος στα συστήματα μου, είναι απολύτως ασφαλή. Πάντα έχουμε καθυστέρηση έναντι όλων αυτών των επιθέσεων, καθότι όλος αυτός ο ψηφιακός κόσμος, οι ψηφιακές τεχνολογίες έφτασαν σε μας χωρίς να έχουμε επίγνωση των ε, απειλών και των ε, προβλημάτων που τους συνοδεύουν. Τώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις των κρατών μελών, εγώ μπορώ να μιλήσω για τη δική μου χώρα, τη Γαλλία. Εδώ και λίγα χρόνια, από το 2009 δηλαδή, ιδρύθηκε η υπηρεσία την οποία διευθύνω και από τότε μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί σημαντικές αποφάσεις για την προστασία των συστημάτων ζωτικής σημασίας και στον τομέα της άμυνας αλλά και σε άλλους οικονομικούς τομείς με σκοπό τα θέματα ασφάλειας του κυβέρνου χώρου να ληφθούν υπόψη σαν μια εθνική προτεραιότητα. Τα μέσα που διαθέτουμε είναι σημαντικά, λοιπόν, ιδιαίτερα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης. Είμαι ένας από τους λίγους διευθυντές τέτοιες υπηρεσίες που, ε, αν και τα κονδύλια που διαθέτω δεν αρκούν, δεν έχω ε, παράπονα όσον αφορά τη χρηματοδότηση του οργανισμού μου. Και βεβαίως για την προστασία των ζωτική σημασίας υποδομών πρέπει να περάσουμε από νομοθεσία για να υπάρξει αποτελεσματική προστασία, το οποίο ε, προϋποθέτει περισσότερο χρόνο. Θα επανέλθω σε αυτό που είπατε όσον αφορά τον προστατευτισμό. Δεν είναι δική μου δουλειά αυτή. Η δική μου δουλειά είναι η ασφάλεια. Και η ασφάλεια προϋποθέτει εμπιστοσύνη στον εξοπλισμό, στους φορείς παροχής υπηρεσιών και σε όλα τα οικοσυστήματα στα οποία λειτουργούμε. Αυτό που είπα και μπορεί να εκλειφθεί ενδεχομένω σαν προστατευτισμός είναι η εμπιστοσύνη προέρχεται από τη γνώση. Πρέπει να γνωρίζω το περιεχόμενο των συστημάτων. Άρα η κρυπτογράφηση προϋποθέτει κάποιες γνώσεις πιο συγκεκριμένες. Δεν μπορώ να κοιτάω μόνο το περιτύλιγμα, πρέπει να μπω στο περιεχόμενο. Για να μπορέσω να το πιστοποιήσω, να ξέρω αν είναι ένα σύστημα ασφαλές. Πολλές φορές λοιπόν δεν ε, πρόκειται για ευρωπαϊκά συστήματα. Χρειάζομαι όμως να έχω τον κωδικό, να μπορώ να διεισδύσω και να γνωρίζω καλύτερα περί τίνος πρόκειται. Και βεβαίως κάθε φορά που αναφερόμαστε σε συστήματα που αφορούν αυτή την αποκρυπτογράφηση θα πρέπει να μπορούμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα όλων αυτών των συστημάτων, των φορέων παροχής υπηρεσιών και αν κάποιος θέλει με τοπικές ρυθμίσεις να προστατευθεί θα πρέπει να επιβάλλει την αποθήκευση όλων αυτών των δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το έχουμε ήδη επιβάλει στη Γαλλία και βεβαίως δεν μιλάμε για e-cloud, μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο μας επιτρέπει να ελέγχουμε το επίπεδο ασφάλειας ε, που προσφέρουν αυτοί οι φορείς ε, παροχής υπηρεσιών στην Ευρώπη. Τουλάχιστον στη Γαλλία δεν απαγορεύουμε σε κανέναν επιχειρηματία εκτός Ευρώπης να λάβει την πιστοποίηση βάσει των κανόνων που έχουμε καθορίσει εμείς όμως στην Ευρώπη. Και όλα αυτά βεβαίως εξαρτώνται από την ε, εμπιστοσύνη που μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα συστήματα και γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να μπορούμε να δυσδύσουμε και να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Βεβαίως συνεργαζόμαστε με τους ε, συναδέλφους από το κέντρο του ΝΑΤΟ στην Εστονία. Και αυτή η συνεργασία είναι πολύ σημαντική και στο θέμα της συνεργασίας αυτής καθεαυτής, αλλά όχι μόνο στον τομέα της άμυνας, Πολλές από αυτές τις ε, τεχνολογίες δεν αφορούν μόνο τον αμυντικό τομέα και βεβαίως ε, το ΝΑΤΟ μας προστατεύει κατά αυτών των στρατηγικών απειλών. Οι σύμμαχοί μας ενδιαφέρονται για τις τεχνολογίες που διαθέτουμε, για τα δίκτυά μας και δεν μπορούμε πάντα να βασιστούμε στους εταίρους μας όσον αφορά την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής που διαθέτουμε. Πρέπει να κινητοποιήσουμε όλους τους φορείς, τους πολίτες. Αυτός είναι ένας τρόπος προστασίας και η περίπτωση της Εστονίας ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερη. Η λειτουργία των Cyber Leagues παραδείγματο χάρη, είναι κάτι το ιδιαίτερο για την Εστονία και δεν νομίζω ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλε χώρε. Εμεί όμω βασιστήκαμε σε αυτό το μοντέλο, εμπνευστήκαμε και δημιουργήσαμε ένα είδους ε, αποθεματικού θα έλεγα, γιατί σε περίπτωση επίθεσης ξέρουμε ότι σίγουρα θα χρειαστούμε άτομα που με μεγάλη ταχύτητα θα μπορέσουν να ξαναδημιουργήσουν δίκτυα. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με το Υπουργείο Άμυνας και θέλουμε να έχουμε άτομα διαθέσιμα, περίπου χίλια άτομα διαθέσιμα, τα οποία σε περίπτωση ανάγκης να μπορέσουν να δράσουν με ταχύτητα και να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των δικτύων. Άτομα τα οποία θα μπορέσουν να δράσουν και να βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των δικτύων. Τώρα, αναφερθήκατε στα βήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Σίγουρα σε πολλά κράτη-μέλη θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η λειτουργία βάσει δικτύων, βάσει εμπιστοσύνης. Θα πρέπει να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό πιστεύουμε ότι σιγά σιγά θα γίνει. Όμως σε κάθε περίπτωση μη λήψη υπόψη των προβλημάτων ασφάλειας στο σωστό επίπεδο, σίγουρα θα δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Θα θεωρήσει κανείς καταρχήν ότι πρόκειται είτε για δυναμία είτε για ε, αδιαφορία των ε, ηγετών, αυτών που θα έπρεπε να λάβουν κάποιες ε, πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις. Προς το παρόν τα θύματα αντιμετωπίζονται σαν θύματα, όμως πολύ σύντομα αυτοί οι οποίοι δεν υλοποιούν τις ρυθμίσεις, τους κανονισμούς, δεν εφαρμόζουν την νομοθεσία, αυτοί που δεν λαμβάνουν τα μέτρα για την προστασία τους σίγουρα θα θεωρηθούν πολύ σύντομα υπεύθυνοι. Ολοκληρώνω και το σήμερα, νομίζω το παρουσιάσατε εσείς, μιλήσατε για την οδηγία νης και την δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη. Η αξιολόγηση των συστημάτων, των προϊόντων, των φορέων παροχής υπηρεσιών, η πιστοποίηση σίγουρα θα δημιουργήσει περισσότερη εμπιστοσύνη. Χρειαζόμαστε προτεραιότητες και εμείς στη Γαλλία έχουμε θέσει κάποιες προτεραιότητες, δηλαδή τα διάφορα δίκτυα ερωτικής σημασίας, τα μεγάλα δίκτυα των κρατών μελών, τα μεγάλα διευρωπαϊκά δίκτυα, αλλά και μικρότερη στόχοι. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι ανησυχώ ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις με δέκα υπαλλήλου, παραδείγματο χάρη, που δεν μπορούν από μόνοι τους να διαχειριστούν την ασφάλεια των συστημάτων τους, το αναθέτουν λοιπόν σε εξωτερικούς φορείς. Γι' αυτό και όλες αυτές οι λύσεις που θα μπορούν να είναι εύχριστες ε, και μέσω cloud computing αλλά και μέσω άλλων τεχνολογιών που να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εύκολα να χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να στηριχθούν από εμάς με σκοπό την οικοδόμηση περισσότερης εμπιστοσύνης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πουπάρ για την παρουσίασή σας και για τον τρόπο με τον οποίο λάβει χώρα διάλογό σας με τα μέλη. Αναφερθήκατε και στο νομοθετικό έργο κατά τη διάρκεια της παρουσίασης θα δώσουμε συνέχεια σε αυτό με τα μέλη και θα το συζητήσουμε τους συντονιστές, να δούμε τι συνέχεια μπορούμε να δώσουμε όσον αφορά την ασφάλεια στον τομέα αυτό στην Ευρώπη. Πιθανότατα θα γίνει και κάποια διάσκεψη πάνω σε αυτό. Διάσκεψη ψηλού επίπεδου. Θα είμαστε σε επαφή μαζί σα και θα σα ενημερώσουμε δεόντω. Ευχαριστώ και εσάς και τα μέλη για τι έξοχες ερωτήσει του. Σα ευχαριστώ. Συνάδελφοι, πάμε στο σημείο 5 Ευρωπαϊκό Ταξιδιωτικό Έγγραφο για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκών τρίτων χωρών. Διαδικαστικό. Ναι. Πριν πάμε στο επόμενο σημείο, αυτή η ανταλλαγή απόψεων έλαβε χώρα στα πλαίσια της συνέχειας που δίδεται στην έρευνα που διεξήχθη. Εγώ ανέφερα την υπόθεση Belgacom. Είναι αξιοσημείωτο, ξοδεύουμε πολύ χρόνο εμείς συζητώντα το θέμα αλλά μπήκε στο αρχείο η υπόθεση και φαίνεται την ξεχάσαμε κι εμείς. Μπορούμε να επανέλθουμε και σε αυτό. Μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβη. Διότι η Foxit, η εταιρεία που ερεύνησε την υπόθεση, άρχισε να ανακαλύπτει κάποια πράγματα. Έφνης, ανεξήγητα, την απέσυραν από την υπόθεση. Και τώρα η δικαστική έρευνα σταμάτησε. Διότι δεν ευρέθησαν αποδείξεις. Θα ήταν ενδιαφέρον να καλέσουμε κάποιους από τους ομιλητές να επανέλθουν κυρίως υπευθύνους της Foxit και να μας εξηγήσουν περίπου τι συνέβη. Καλώς κύριε Ντφέλτ, θα το θέσω στους συντονιστές. Ακολουθεί συνεδρία των συντονιστών σήμερα. Αυτή η συζήτηση δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς να αναφέρουμε την υπόθεση Belgacom. Σας ευχαριστούμε. Εντάξει, εσείς συγχωρήστε, μπορείτε να αποχωρήσετε. Ευχαριστώ. Όπως έλεγα, πήγαμε στο σημείο 5 παρουσίαση του τριμερούς διαλόγου που βρίσκονται συζητήσεις. Θα μας ενημερώσει ο κύριος Χαλοάχο για το θέμα αυτό. Ο κύριος Χαλοάχο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό σε ένα τεχνικό και ένα πολιτικό τριμερή διάλογο. Είναι πολύ σημαντικό για το σύστημα ασύλου μας να διασφαλίσουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των εγγράφων και των τεχνικών διαδικασιών που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να συνεργαστεί με ευρωπαϊκές χώρες. Η συμφωνία αυτή ελπίζουμε ότι βελτίωσε τα ταξιδιωτικά μας έγγραφα για το μέλλον. Έχουμε ένα έγγραφο το οποίο χρησιμοποιείται όλο ένα και περισσότερο από τα κράτη-μέλη και θα αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο από το τρίτες χώρες. Οι βασικές αλλαγές στην αρχική πρόταση περιλαμβάνουν τα εξής. Στην ε, αιτιολογική σκέψη παριθμών 7, το Κοινοβούλιο κατάφερε να παραμείνει η αναφορά στην επανεισδοχή και την ανάγκη της αναγνώρισης του ταξιδιωτικού εγγράφου, το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στι διαπραγματεύσεις με τους διπλωματικούς εκπροσώπους τρίτων χωρών όταν συζητούνται ε, οι αποστολέ αυτέ. Στην αιτιολογική σκέψη 22 το Κοινοβούλιο διατήρησε την αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών με άση της αναφοράς στο άρθρο 39 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την ανάγκη να σεβόμαστε διεθνείς και ευρωπαϊκές ε, νομικές υποχρεώσει. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό προς το Κοινοβούλιο οι επιστροφές και το θέμα των ε, ταξιδιωτικών εγγράφων να περιλαμβάνονται ε, στο υπόλοιπο ε, κεκτημένο για το άσυλο. Το άρθρο 3, παράγραφος 3, αναφέρεται σε ένα ταξιδιωτικό έγγραφο το οποίο ισχύει για ένα ταξίδι μέχρι να έχει φτάσει ο υπήκο τρίτη χώρας στη χώρα προορισμού του. Ε, αυτό ε, μπορεί να ε, βοηθήσει για πιθανές δυσκολίες στο ταξίδι πριν φτάσει στον προορισμό του. Επίσης, μας ενδιαφέρει να εγκατοπτρίζεται και το σκεπτικό μα για τι πράξει κατεξουσιοδότηση βάσει τη Διοργανική συμφωνία για την καλύτερη νομοθεσία. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, συμφωνίας ήταν να διασφαλίσουμε ε, πλήρη αναθεώρηση του εγγράφου το αργότερο τρεις μήνες ε, μετά από την έναρξη ισχύω, παρά την προβλεπόμενη διαδικασία αναθεώρησης. Μετά από αυτό το έγγραφο θα συμπεριληφθεί στην αναθεώρηση της οδηγίας για τις επιστροφές. Αυτό θα είναι το νέο άρθρο 8 είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσουν ότι δεν θα περιμένουμε χρόνια πριν ε, αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτού του αναθεωρημένου ταξιδιωτικού εγγράφου και ε, να κάνουμε και κατάλληλες αλλαγές αν χρειαστεί. Επίση, δεν υπάρχει καμία αναφορά στο τελικό κείμενο στην ανταλλαγή των πληροφοριών και την αποθήκευση των πληροφοριών στις βάσεις δεδομένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. είναι κατανοητό ότι τα θέματα αυτά θα τα συζητήσουμε στο μέλλον σε ξεχωριστό μέσο. Το άρθρο 9 ζητά το έγγραφο αυτό να εφαρμόζεται τέσσερις μήνες μετά την ε, θέση σε ισχύ του κανονισμού αυτού για να επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να προσαρμοστούν με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται και να προσαρμόσουν και τα σχετικά συστήματα πληροφορική τους. Το άρθρο 12 που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου Προβλέπει επίσης και πιθανές μελλοντικές ε, εξελίξεις ε, στα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τις τεχνικές προδιαγραφές. Όπως σας έχω πει και στο παρελθόν, αυτό το ταξιδιωτικό έγγραφο δεν αποτελεί μαγική λύση για τα προβλήματα για τη μετανάστευση ή τα προβλήματα που έχουμε σε θέματα επιστροφών. Αλλά είναι ένα τμήμα του μοσαϊκού και είναι και ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Επικαιροποιώντας τα, τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, το οδεύουμε προς ένα σύστημα ασύλου το οποίο θα είναι καλύτερο και θα είναι καλύτερα εξοπλισμένο να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτή τη στιγμή ένα βασικό πρώτη με τις πρόκλησεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι να έχουμε ένα αποτελεσματικό τρόπο επιστροφών. Όπως μάθαμε, λιγότερες από τις μισές αποφάσεις επιστροφών εφαρμόζονται. Επομένως, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ολλανδική Προεδρία, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους κοιόδης συγητέ για τη συνεργασία τους και την αποτελεσματική ε, δουλειά τους και ελπίζω να υποστηρίξετε όλοι αύριο τα αποτελέσματα στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος το λόγο από τους κοιόδης συγητές. Όχι. Αν όχι, η ψηφοφορία για την πολιτική συμφωνία θα γίνει αύριο στην Επιτροπή μας και ψηφοφορία στην Ολομέλεια το Σεπτέμβριο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χαλάχο. Περνάμε τώρα στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που είναι παρουσίαση από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Φόρουμ Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του 2016 έγινε στη Βιέννη 20 με 23 Ιουνίου του 2016. Ήταν μια εκδήλωση στην οποία είχαμε ηθήνοντες, ε, ενδιαφερομένους για να αντιμετωπίσουμε και να συζητήσουμε τις προκλήσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είχαμε και πολλούς ε, ευρωβουλευτές και μέλη της Επιτροπής μας ε, που συμμετείχαν στις εργασίες. Σήμερα είναι εδώ ο κύριος, ε, η κυρία συγγνώμη, Τζοάννα Γκούντι, προϊστάμενη του Τμήματος Ελευθεριών και Δικαιοσύνης, για να μας παρουσιάσει τα αποτελέσματα του φόρουμ και τις δηλώσεις που αποφασίστηκαν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΛΥΜΠΕ και τη ΛΥΜΠΕ που με κάλεσαν εδώ σήμερα να μιλήσω εκ μέρους του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, να σας ενημερώσω περί των αποτελεσμάτων της ευρύτερης για μας ε, μέχρι τώρα διάσκεψης, το Φόρουμ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, με άλλα λόγια. Αν μέτρησα σωστά, 10 ευρωβουλευτές και αρκετοί από τους παριστάμενους συμμετείχαν στο φόρουμ αυτό και σας ευχαριστώ πολύ για την ενεργό συμμετοχή σας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία του φόρουμ. Είχαμε τον τίτλο «Ευρώπη των αξιών στο σημερινό κόσμο» σαν τίτλο του φόρουμ. Ο διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, Michael O'Flaherty, έθεσε το θέμα ως συζήτηση θεμελιώδη δικαιώματα περίοδο κρίσης. Πάνω από 700 ήταν οι συμμετέχοντες και κάποιοι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά κυρίω ήταν οι εκπρόσωποι των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεως. Εκπροσωπήθηκαμε σε ύψιστο επίπεδο τον πρώτο αντιπρόεδρο, τον κ. Τίμερμανς, ο οποίο άνοιξε τη διάσκεψη. Είχαμε εκπροσωπού από Ιρλανδία, Πολωνία, Σλοβακία και πολλού υψηλού αξιωματούχου αξιωματούχους από αρκετά άλλα κράτη-μέλη που αυτό έδειχνε το υψηλό ενδιαφέρον από εκείνους που υπέχουν το καθήκον και εκτελούν το καθήκον αυτό. Είχαμε υψηλή εκπροσώπηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίπεδο Γενικών Διευθυντών, είχαμε κάποιου ευρωβουλευτέ, και υψηλού εξωματούχου των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπη. Αυτό που θέλω να τονίσω επίσης είναι και κάτι εξίσου σημαντικό, ότι είχαμε εκπροσώπους από πολλούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ, εκπροσώπους επιχειρηματικού, του επιχειρηματικού κόσμου, πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους των τεχνών, όλοι εκπροσωπήθηκαν στο φόρουμ αυτό. Το φόρουμ διοργανώθηκε πάνω σε τρία βασικά θέματα δεν είχαμε τη συνηθισμένη προσέγγιση προηγουμένων διασκέψεων με ένα θέμα. Εδώ είχαμε τρία θέματα. Τα εξή. Προστασία των προσφύγων το πρώτο θέμα. Βέβαια έπρεπε να ασχοληθούμε με το θέμα προστασία των προσφύγων. Ήταν η μεγαλύτερη κρίση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερο ζήτημα ήταν η συμπερίληψη, ένταξη Έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές κοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται ισότητα και δικαιώματα για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτο θέμα, είχαμε το νέο πρόβλημα να καλύψουμε όλα αυτά τα ζητήματα, να δημιουργούνται, δημιουργούνται ευκαιρίες αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά υπάρχουν και απειλές που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αυτά ήταν τα τρία βασικά θέματα, συζητήθηκαν από πάνελ, έγιναν παρουσιάσεις, και γίνηκαν διάφορε ομιλίε προ προβληματισμό και δημιουργήσαμε 28 παράλληλε ομάδε εργασία. Ποια ήταν βασικά αποτελέσματα, η δήλωση του Προέδρου. Τι δηλώσει έχετε εδώ, στο τραπέζι. Ένα λεπτό έγγραφο είναι, αλλά είναι πληρέστατο. Να παρουσιάσω εν συντομία κάποια βασικά σημεία των δηλώσεων του Προέδρου. Ο Προέδρος του Φόρουμ ήταν διευθυντή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο Μάικλ Οφλάερτη αλλά η δήλωση του Προέδρου δεν αποτελεί αποκλειστική δική του δήλωση, προσπαθεί να α, δείξει ποιο ήταν το πνεύμα όλων των εργαζομένων στη διάσκεψη. Δεν είναι ένα συμπεφωνημένο κείμενο, δεν δεσμεύονται οι συμμετέχοντες και συγκεκριμένες δράσεις, όμως περιγράφονται βασικοί τομείς που τονίστηκαν στη συζήτηση του φόρουμ. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν ποιες δράσεις θεωρούν απαραίτητες. Στη δήλωση προσπαθούμε να ε, διηλύσουμε όλα αυτά και να απευθυνθούμε προς τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και άλλους φορείς, όπως είναι φορείς του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών, να τους δείξουμε ποιοι τομείς χρήζουν δράσεως όταν μιλάμε για θεμελιώδη δικαιώματα σε περίοδο κρίσεως. Ποιε είναι οι βασικέ προτάσει προ δράση, αυτέ που περιγράφονται στη δηλώση του Προέδρου. Πρώτο θέμα προστασία προσφύγων. Τονίζεται όλος ιδιαίτερα η βασική ανάγκη χρήσεων προδιαγραφών τα ανθρώπινα δικαιώματα που θα κατευθύνουν τι πολιτικές περί προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό όσον αφορά τις απαιτούμενε δράσεις. Οι συμμετέχοντες ζήτησαν πρακτικά μέτρα από πλευρά θεσμικών οργάνων και κρατών μελών. Επί παραδείγματι, να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να εντοπιστούν όλα τα εργαλεία και μέτρα για να μην έχουμε στέρηση ελευθεριών των ετούντων ασύλων. Κάτι άλλο. Πρέπει να εγγυηθούμε την προστασία των ευάλωτων ομάδων, όπως ασυνόδευτα παιδιά. Πρέπει να εξαιρούνται από επιταχυμένες διαδικασίες για τη χορήγηση ασύλου. Μετά, ο αντίκτυπος της κρίσης των προσφύγων στις τοπικές κοινότητες. Ακούστε και πρακτική σύσταση που είναι και στη δήλωση του Προέδρου. Δηλαδή τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα για να αντισταθμίσουν τα προβλήματα των τοπικών κοινοτήτων όταν υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα από την κρίση. Αναγνωρίζεται η κοινωνική και η οικονομική θέση αυτών των ομάδων. Παραδείγματο χάρη, όταν έχει καταρρεύσει ο τοπικό πληθυσμό. Για κάθε ευρώ που δαπανάτε, προτάθηκε, για κάθε ευρώ που δαπανάτε τι πρόσφυγε, ένα ευρώ θα μπορούσε να απανηθεί για τον τόπιο πληθυσμό και τι ντόπιε υποδομέ. Και εδώ η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συνεργαστεί με την κοινωνία των πολιτών και τι τοπικέ επιχειρήσει Κάτι άλλο τονίστηκε. Η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστασία των αφιχθέντων. Πολλοί από εκείνους που αφικνούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από περιοχές συγκρούσεων υποφέρουν από τραύμα, από σοβαρά προβλήματα. Θα πρέπει ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και, εθνική, ε, και τα εθνικά συστήματα υγείας να στηρίξουν ψυχολογικά αυτά τα άτομα και να τους δοθούν και συμβουλές. Και κάτι τέτοιο δεν κοστίζει ακριβά. Το θέμα νέας τεχνολογίας για όλους, για να ανταποκριθούν στην κρίση, ήταν ένα σημαντικό θέμα που τονίστηκε. Κάτι πολύ σημαντικό. Προστασία των παιδιών που μετακινούνται. Εκεί χρειάζεται δράση. Αυτό αναφέρθηκε στο φόρουμ. Δηλώθηκε ότι συστήματα προστασίας πρέπει να προωθούν τα καλύτερα συμφέροντα των παιδιών. Αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο των δράσεων. Π.χ. ταυτοποίηση και καταχώρηση όλων των ασυνοδεύτων παιδιών. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί χρησιμοποιώντα μέσα κατάρτιση για αυτού που ασχολούνται με το θέμα. Τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τα κράτη-μέλη μπορεί να βοηθήσουν. Να υπάρχει συστηματική κατάρτιση για προστασία των παιδιών και τα δικαιώματα των παιδιών. Να χορηγείται αυτή η κατάρτιση στου διάφορου αρμοδίου. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα στον αυτή την προστασία των προσφύγων. Στρέφουμε προ το δεύτερο βασικό θέμα του φόρουμ. Η ένταξη, η συμπερίληψη. Πολλοί εξέφρασαν ησυχίε. Πρέπει να παρέχονται ίσες ευκαιρίες σε όλους. Αυτό αναφέρθηκε αναγνωρίζοντας το κοινωνικό και πολιτικό κλίμα, το οποίο ανέχεται όλο και περισσότερο εξτρεμισμό, ρατσισμό και ξενοφοβία, που όλα αυτά βασίζονται στους φόβους για την ασφάλεια και την απασχόληση. Λοιπόν, τα κράτη-μέλη πρέπει να ενισχύσουν τους φορείς ισότητας και να προβλέπουν κυρώσεις όταν διαπιστώνεται διάκριση, αποτελεσματικές, αναλόγες και αποτρεπτικές κυρώσεις. Και σε επίπεδο του Διεθνούς Δικαίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αναφέρθηκε η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες, που είναι αναπόσπαστο τμήμα τη ενόμου τάξη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Και είπαμε ότι τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα εκείνων των κρατών μελών που έχουν παράσχει επαρκείς πόρους για να καλύπτονται τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία στην πράξη. Ένα από τα βασικότερα θέματα που διαπιστώθηκε ήταν η παιδεία. Η παιδεία είναι ζωτική σημασία. Ούτω ώστε να έχουμε υπεύθυνου πολίτε που θα στερνίζονται τι κοινέ αξίε όπω την μη διακριτική μεταχείριση. Προτάθηκε κάτι. Ότι οι φορεί επαγγελματική διαπίστευση θα παρέχουν κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους αρμοδίους. Πρέπει τα κοινωνικά δικαιώματα να προωθούνται για πιο ε, δεκτικές κοινωνίες και τα δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να γίνονται σεβαστά. Θα πρέπει να αυξήσουμε και τα ποσοστά απασχολησιμότητας. Τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ενώση και τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τι επιχειρήσει και, τις και την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να βρουν τρόπου για την καταπολέμηση φαινομένων όπως είναι η εκμετάλλευση των εργαζομένων. Το τρίτο θέμα. Ψηφιακή εποχή. Οι άνθρωποι διασυνδέονται μεταξύ τους και επαγγελματικά και σε ιδιωτικό επίπεδο. Και θα πρέπει όμως και στο διαδίκτυο και εκτός διαδικτύου ότι σεβαστά ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή η εποχή μας δίνει ευκαιρίες και απειλές όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το ψηφιακό θεματολόγιο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω είναι αποτελεσματικό εργαλείο για να αποφευθεί ο κοινωνικό αποκλεισμό. Για να ξέρουν καλύτερα τα δικαιώματά του οι άνθρωποι. Προτάθηκε μια ιδέα. Να υπάρχει πρόσβαση σε μηχανισμούς αποζημιώσεως μέσω διαφόρων εφαρμογών ψηφιακών, ούτω ώστε και πλέον απόμακρες περιοχές να καλύπτονται. Νέες τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλεία κατά των καταχρήσεων και κακομεταχείρισης. Μίσος που εκφράζεται μέσω διαδικτύου γίνεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και αν δεν αντιμετωπιστεί αυτό θα αυξηθεί σαν φαινόμενο. Τα δικαιώματα και οι ευθύνες θα πρέπει να προωθούνται στην ψηφιακή εποχή. Έχουμε και ένα πακέτο για την προστασία των δεδομένων. Πρέπει να προωθηθεί. Προτάθηκαν και διάφορες πρακτικές πρωτοβουλίε όσον αφορά την ψυχιακή εποχή. Να παραθέσω κάποια παραδείγματα. Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων μέσω νέων εφαρμογών στον τομέα τη ηλεκτρονική υγεία. Αυτό απαιτεί μέτρα διαφύλαξη για τα προσωπικά δεδομένα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό όσον αφορά τη διαχείριση των στοιχείων. Διότι ανατίθεται η διαχείριση των δεδομένων στον ιδιωτικό τομέα και περισσότερο. Κοινά μαθήματα στα πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα απαιτείται να γίνει. Εκεί που μελετώνται ε, μελετείται ο νόμος, αν θέλετε. Ασχολούνται με τη νομική. Και θα πρέπει επίσης να σχεδιάζονται κατάλληλα και μελλοντικέ εφαρμογές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλη πρακτική πρόταση. Ένα σύστημα που θα χρησιμοποιεί ψυχιακή τεχνολογία που θα χρησιμοποιούν οι εταιρείε με τις ρυθμιστικού φορείς δηλαδή κόκκινο, πράσινο, κίτρινο φως Δηλαδή, αν υπάρχει σύστημα προειδοποίηση κόκκινο, τι σημαίνει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή στο διαδίκτυο και προσωπικά δεδομένα μπορεί να απολυθούν, να ξαναχρησιμοποιηθούν. Άρα πρόσεχε σημαίνει το κόκκινο. Αυτές ήταν κάποιες από τις προτάσεις που ανέφερα. Στο έγγραφο που ανέφερα αναφέρονται λύσεις για τα προβλήματα. Και στα απορίσματα των 28 ομάδων εργασίας αναφέρονται λεπτομέρειες. Θα βρείτε στο διαδίκτυο σύντομα τα πορίσματα των ομάδων εργασία. Ο Πρόεδρο αναφέρεται στου διάφορου φορεί και εκείνου που είναι υπεύθυνοι. Πώ μπορούν να προωθήσουν τη συμμόρφωση των τα ανθρώπινα δικαιώματα στου τρεις που αναφερθέντες τομείς. Αναφέρεται επίση ο οργανισμό μα τι θα κάνει. στι σελίδε 36 έω 40 στι δηλώσει του Προέδρου αναφέρεται τι θα κάνει ο οργανισμό μας. Λοιπόν, Αναφέρεται επίσης η αναγνώριση των σχέσεων μεταξύ τομέων και φορέων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα κράτη-μέλη, οι αρχέ των κρατών μελών, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η κοινωνία των πολιτών, οι διεθνεί οργανισμοί, ο επιχειρηματικό τομέα, τα πανεπιστήμια που παρίστανται στο φόρουμ, αν συνεργαστούν όλοι αυτοί, μπορούν να προωθήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα για όλου. Έδειξε το φόρουμ ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε διάφορες πτυχές δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να δούμε και πέρα από το παραδοσιακό μας ακροατήριο τα ανθρώπινα δικαιώματα Στη σελίδα 3 και 4 των, της δηλώσεως των Προέδρων βλέπετε τέσσερα βασικά θέματα του φόρουμ. Πέρα από τους βασικούς τομείς, τους θεματικούς, είχαμε και άλλους τέσσερις τομείς που διαφάνησαν. Σας αναφέρω ακροθυγός. Πρώτον, τα θεμελιώδη δικαιώματα εφαρμόζουν τη σπάση σωστά εστιαστήκαμε επί συγκεκριμένων ομάδων κοινωνικών, που είναι ευάλωτε ομάδε. Και είπαμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να καλύπτουν πάντε στου πάντες. Η αναφορά στην ψηφιακή εποχή είναι σαφέστατη. Προωθεί η ψυχιακή εποχή τα δικαιώματα, αλλά δημιουργούνται και απειλέ. Ένταξη. Όλοι πρέπει να εντάσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να καλύπτονται και οι νέοι και οι ηλικιωμένοι στον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και διαφορετικά άτομα. Δεύτερο θέμα. Παιδεία. Παιδεία περί θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πολύ σημαντική σε διάφορα επίπεδα. Φερρυπίν. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι πανεπιστήμιο. Από τον ιδιωτικό τομέα μέχρι το δημόσιο τομέα. Κατάρτιση. Επίσης δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η εκπαίδευση στα θεμελιώδη δικαιώματα χρησιμοποιήσει νέα γλώσσα για να αυξηθεί η προσβασιμότητα σε αυτά. Τρίτο γενικό σημείο. θεσμική λογοδοσία. Αν υπάρχουν παραβιάσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, αυτό πρέπει να διώκεται. Τέταρτον, για τα άτομα με αναπηρίες. Τίποτα που μας περιβάλλει δεν μπορεί να είναι χωρίς εμάς πρέπει να εφαρμοστεί για τα θεμελιώδη δικαιώματα, για τα άτομα με αναπηρία. Τίποτα που μα αφορά χωρί εμά, Άρα χρειάζεται συνεργασία εκείνων που προβληματίζονται, που έχουν το πρόβλημα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματά του, τα θεμελιώδη δικαιώματά του και να του λαμβάνουμε υπόψη όταν θεσπίσουμε νομοθεσία. Ο Οργανισμός Θεμελιώδη Δικαιώματα θα αναφερθεί στι 100 πρακτικέ προτάσει που αναφέρονται στι δηλώσει του Προέδρου. Θα τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά στι εργασίε μα. Ελπίζουμε ότι εσείς, σαν Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, μπορείτε να αναφερθείτε σε αυτά που συστήνει ο Πρόεδρος και να συνεργαστείτε μαζί μας. Και έτσι και το επόμενο φόρουμ να είναι πολύ καλή εκδήλωση και να είναι επιτυχής εκδήλωση. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Ευχαριστώ συνάδελφοι, όλοι έχετε αυτό το βιβλιαράκι. Κάποιοι από εσάς ήσασταν παρόντες. Μόνο μέχρι τις 16.45 έχουμε. Πριν έχουμε το θέμα της προστασίας ιδιωτικότητας και μετά έχουμε και κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΕΚΟΝ. Τέταρτο έχουμε στη διάθεσή μας. Δύο συνάδελφοι είναι στον κατάλογο μιλητών. Ποιος άλλος θέλει. Όλοι να μου πείτε τώρα αν θέλετε να μιλήσετε. Και Άννα. Πείτε το μου τώρα, σηκώστε το χέρι. Θέλετε να μιλήσετε ή όχι. Ωραία. Κανείς άλλος. Πολύ σύντομη να είστε. Δεν θα έχετε ώρα να απαντήσετε βέβαια. Είχαμε μισή ώρα για το θέμα, βλέπετε. Εντάξει, τους γράψατε όλους. Ωραία. Τέλεια. Δεν ξέρω. Um, we Μπόνι, ευχαριστώ πολύ. Εγώ συμμετείχα στο φόρουμ κατά την ημέρα που επικεντρωθήκαμε στην ψηφιακή εποχή και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια πολύ καλά οργανωμένη συζήτηση, διότι θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα και ήταν μια ευκαιρία να συναντήσουμε αρκετούς ε, ε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλους και ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ σε κάποια σημεία. Πρώτον, η αναγνώριση ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου εντό και εκτό διαδικτύου. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίση, αναφέρθηκε ότι στη διάρκεια τη εφαρμογή ε, του ε, νομοθεσίας θα πρέπει να γίνει από κοινού, από όλα τα θεσμικά όργανα, από όλα τα επίπεδα, από όλους τους και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τρίτον, Πρέπει να το σκεφτούμε, ήταν και πρόταση αυτό, ε, κάποια χάρτα δικαιωμάτων που θα αφορά τη ε, προβλήματα που υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Ήταν μία εκ των προτάσεων του φόρουμ αυτή και νομίζω ότι ακούστηκε με ιδιαίτερα στένος το γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο οι επιχειρήσεις και όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεργαστούν με οργανώσεις ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε αυτή την πρόταση η οποία αφορά αυτό το σύστημα του φωτεινού σηματοδότη για τους χρήστες της ψηφιακής τεχνολογίας και Ακούστηκε αυτό και στη διάρκεια της ε, ε, συζήτησης. Θα πρέπει να συζητήσουμε με επιχειρήσεις αλλά και με ρυθμιστικές αρχές. Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διάσκεψη. Ευχαριστώ η κυρία Λόριστετ. Ευχαριστώ πολύ. να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Μπόνι. Και εμείς ήμασταν, και εγώ ήμουν εκεί στη συζήτηση για την ψηφιακή εποχή και πρέπει να πω ότι πολύ συχνά αυτές οι εκδηλώσεις τείνουν να είναι πολύ επίσημες και τελετουργικές και ήταν θετική έκπληξη για μένα το γεγονός ότι η ατμόσφαιρα στη διάρκεια της συνεδρίας ήταν πάρα πολύ σοβαρή και υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή και οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι συζήτησαν ανοιχτά τα διάφορα ζητήματα. Κατ' εμέ, ένα από τα ουσιαστικά ζητήματα τα οποία επαναλαμβάνονταν συνεχώς είναι ότι πρέπει να εξετάσουμε την παιδεία ε, στην ψηφιακή εποχή πάρα πολύ σοβαρά και ε, να ε, δούμε την εκπαίδευση και την τεχνολογία σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι αναφερόμαστε στην προστασία του, της προσωπικής ζωής ε, ε, αλλά εάν δεν υπάρχουν άνθρωποι που δεν αντιλαμβάνονται την εκπαίδευση και την τεχνολογία θα έχουμε προβλήματα στην εφαρμογή μετά. Κάτι άλλο το οποίο ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικό και λήφθη πολύ σοβαρά υπόψη είναι το θέμα της ε, ένταξης. Αυτή η νέα εποχή εμφανίζεται ως κάτι φυσιολογικό για τους νέους ανθρώπους, αλλά αναφέρθηκε και η γυράσκουσα ε, πλευρά του πληθυσμού ε, και όλοι αυτοί που είναι άνω των 40 θα έλεγα που πρέπει ε, να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους και το θέμα αυτό. Πρέπει να ενταχθούν και αυτοί και να υπάρχει ισότητα και για αυτούς, όχι μόνο για τα άτομα με αναπηρία που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για όλες αυτές τις ομάδες πληθυσμού. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή συζήτηση και ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι περαιτέρω και να το προχωρήσουμε, διότι ήταν πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Ε, ήταν πολύ σημαντική και η δημιουργικότητα, το γεγονό ότι μπορούμε να έχουμε ένα νέο βήμα προ συζήτηση και όλα αυτά. Κύριε Γκόμε, δυστυχώ εγώ δεν μπόρεσα να συμμετέχω. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα μέλη να μπορούν να συμμετέχουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα συμπεράσματα την προστασία και όλα αυτά τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά. διότι ο τομέας αυτός ε, έρχεται σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αξίες της και χάνει αξιοπιστία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες και η ερώτησή μου είναι κατά πόσον σκοπεύετε να κάνετε κάτι, να κάνετε συγκεκριμένη έρευνα και να μας παρουσιάσετε τα συμπεράσματά σας για το κατά πόσον τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά ε, όργανα και υπηρεσίες ζητούν τη συνδρομή σας για να αντιμετωπίσουν προβλήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σε όλα, για παράδειγμα, τους ε, προσφυγικούς καταβλισμούς που έχουμε τώρα στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες ε, καταχρήσεις και κακοποιήσεις ε, για ανηλίκους για παράδειγμα που δεν υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την υπόθεση ενός συγκεκριμένου ανήλικου πρόσφυγα και γυναίκες και παιδιά δεν έχουν βασικά δικαιώματα επανένωση οικογενειών. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ευθύνε όχι μόνο για τι χώρε φιλοξενία, αλλά και για όλου του υπόλοιπου που θα έπρεπε να συνεργάζονται μαζί του. Και υπάρχει και το ψηφιακό χάσμα, το οποίο έχει δημιουργήσει κάποιες πολύ στρεβλές πτυχές. Ε, λέγεται στους πρόσφυγες ότι πρέπει να συνδεθούν μέσω Skype που δεν έχουν γιατί δεν υπάρχει διαθέσιμο Skype και αυτό είναι κάτι το οποίο το προωθούν Ευρωπαίοι υπάλληλοι και υπάλληλοι των χωρών φιλοξενίας. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν για να δώσετε προτεραιότητα στους πρόσφυγες και στα δικαιώματά τους, όπως αναφέρεται αυτό στη δήλωση. Και φυσικά εγώ σας ενθαρρύνω να δράσετε. Ε, συνάδελφοι, μέχρι τις 5 παρατέταρτο, η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Είναι πολύ σημαντικό που το Κοινοβούλιο μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια διοργάνωση και ήταν εξαιρετική. Μας αναφέρατε κάποια από τα αποτελέσματα και εμείς σαν πολιτική ομάδα έχουμε κάποιες ανησυχίες. Όσον αφορά τον κοινωνικό αποκλεισμό και όσον αφορά το θέμα των Ρωμά, η ενσωμάτωση αυτής της ομάδας των Ρωμά βάσει συγκεκριμένων παραμέτρων και δικτών δεν ξέρω αν έχει ληφθεί υπόψη. Το ζητάμε σαν πολιτική ομάδα και θα θέλαμε όσον αφορά την περαιτέρω υλοποίηση της στρατηγικής που αφορά τους Ρωμαία να ενσωματωθεί και αυτό το θέμα στην σειρά των προτεραιοτήτων σας. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Βεβαίως η προβληματική και τα προβλήματα των προσφύγων σήμερα είναι στο προσκήνιο και το θέμα των Ρωμά έχει λίγο ξεχαστεί. Γι' αυτό και θα ήθελα να το αναφέρω. Πολύ σύντομα Θέλω να θέσω κάποιο πρακτικό ζήτημα. Αναφερθήκατε στα 10.000 ε, εξαφανιστέντα παιδιά στην Ευρώπη που είναι παιδιά από οικογένειες μεταναστών και αναφέρθηκε το θέμα στο φόρουμ. Μετά είναι, αναφερθήκαμε και στις δραστηριότητες του οργανισμού. Ζητήσατε πληροφορίες από τη Europol ή από τις αστυνομικές δυνάμεις των ε, κρατών μελών. θα μπορούσαμε να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες για αυτά τα παιδιά. Ε, τι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να χορηγηθούν. Η Σωράγια πώς έχει το λόγο. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την Κορνέλια Ένστ για αυτό που είπε και εκ μέρους των σοσιαλιστών θα ήθελα και εγώ να πω ότι για μας είναι προτεραιότητα η Ρωμά. Κοιτώ την αρχή των ε, προτάσεών σας και βλέπω ότι έχετε συμπεριλάβει δεν βρίσκω αυτό που ήθελα να πω. Θα πάω στη δεύτερη ερώτηση που είχα. Μιλήσατε για τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και η ερώτησή μου είναι εξής. Πώς θέλετε να επεξεργαστείτε αυτό το θέμα στα σχολεία, με καμπάνιες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το θέμα της ξενοφοβίας και το φαινόμενο αυτό δυστυχώς αυξάνεται στην Ευρώπη. Και έχω και μία τρίτη ερώτηση. Εσείς σαν ε, οργανισμός αλλά και εμείς σαν ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ πρέπει να αυξήσουμε τις ε, επαφές μας. Πώς θα μπορούσατε να μας ενημερώνετε περισσότερο. Α, βρήκα αυτό που ήθελα να σας πω προηγουμένως στη σελίδα 5 και 6 το θέμα της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας το διαβάζω αυτό που λέτε, αλλά είναι σαν να λέμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα προστατεύονται βάσει αλληλεγγύης και βάσει αυθαίρετων αποφάσεων. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Και θα ήθελα να μου πείτε συγκεκριμένα τι εννοείτε με αυτή τη φράση. Τώρα, για τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Έχουν το δικαίωμα να ζήσουν με την οικογένειά τους. Και βεβαίως, από τη στιγμή που δεν υπάρχει επανένωση των οικογενειών, αυτό το δικαίωμα παραβιάζεται κατάφορα. Ξέρω βέβαια ότι υπάρχουν ε, οικογένειες ε, που βρίσκουν ε, καταφύγιο στην Σουηδία και άλλες σε μια τρίτη χώρα και δεν θα μπορέσουν ποτέ να επανενωθούν. Πρόεδρος, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Προτείνω για κάποιους που δεν ήταν παρόντες στο φόρουμ ιδιαίτερα. Αν μπορείτε να τους απαντήσετε γραπτά. Ξέρω ότι σημειώσατε όλα αυτά που ρώτησαν τα μέλη της Επιτροπής. Σας το λέω αυτό γιατί περιμένει και ο Επίτροπος ή Επίτροπος. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε για το φόρουμ και για τις ερωτήσεις που υποβάλλεται Ο Οργανισμός για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει μια ευρία εντολή και πολιετές πλαίσιο. Οπότε καλύπτουμε και τους Ρωμά. Είναι από τους εννέα βασικούς τομείς εργασιών μας. Και αναφέρεται και στις δηλώσεις του Προέδρου για την προστασία των προσφύγων. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, μηνιαία εκδίδουμε εκθέσει για την κατάσταση των ετούντων άσυλο σε νέα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω από Σουηδία μέχρι τον Νότο. Πολλά σημαντικά σημεία αναφέρθηκαν όσον αφορά το ψηφιακό χάσμα. Μπορούμε να απαντήσουμε γραπτός, όπως είχε την καλοσύνη να μου πει και ο Πρόεδρος. Έχει εκπνεύσει ο χρόνος μου. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Αυτό που θα κάνουμε είναι να απαντήσουμε γραπτός και να αποστείλουμε τις απαντήσεις στους ευρωβουλευτές. Θα σας δώσουμε τα ονόματα όλων όσων υπέβαλαν ερωτήσει, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Συγγνώμη που έπρεπε να σας διακόψω. Είναι σημαντικό θέμα. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ήθελα να ακούσουμε όλους που ζήτησαν το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Γκούτη. Έξοχη παρουσίασή σας. Συνάδελφοι, Πάμε στο σημείο 7. Ανταλλαγή απόψεων την κυρία Γερόβα για την προστασία των καταναλωτών, Επίτροπο Αρμόδια για τη δικαιοσύνη στους καταναλωτές και της όρθια των φίλων. και περιμένουμε να έρθει εδώ. Um, Θα κάνω την εισαγωγή μέχρι να έρθει. Συνάδελφοι, να υπενθυμίσω σε όλους ότι η Επίτροπος ε, υπέβαλε ένα σχέδιο εκτελεστικής απόφασης που αφορά την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτική Ζωής. Το Κοινοβούλιο ειδοποιήθηκε για αυτή την ε, ε, πρόταση, η οποία είναι βάση του άρθρου 106. Η Επιτροπή ε, ΛΥΜΠΕ συζήτησε το θέμα αυτό τη Δευτέρα 4 Ιουλίου και δεχτήκαμε ευγενικά να ακούσουμε και την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης να σας πω ότι οι συντονιστές θα συναντηθούν αμέσως μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας για να δούνε τι θα κάνουν ε, μετά από τις παρατηρήσεις που θα ακούσουν από την Επίτροπο και η οποία θα απαντήσει και ρωτήσει στην Επιτροπή μας. Θα περιμένω λοιπόν μέχρι να καθίσει η Επίτροπος. If you want to take this time, just indicate. Αν θέλετε εντωμεταξύ να μου πείτε και αν θέλετε να μιλήσετε, ευχαριστώ πολύ. If you want to do that, we can do a complete speaking list and then we can uh, close the list. So if everyone would just indicate now if they want to speak. Να έχουμε ένα πλήρη κατάλογο μιλητών λοιπόν. Σας παρακαλώ πέστε μας αν θέλετε να λάβετε το λόγο στη συνέχεια. Παρακαλώ. Συναδελφοί, έχουμε τρία τέταρτα για αυτή τη συζήτηση. Το λέω και στην Επίτροπο για να ε, φροντίσει να ε, σας αφήσει χρόνο να θέσετε ερωτήσεις και από εκεί και πέρα να μπορέσει να απαντήσει. Όπως ξέρουμε στην Επιτροπή αυτή 45 λεπτά δεν και πολλή ώρα. Έτοιμοι είμαστε εμείς, αν είστε έτοιμοι και εσείς κύριε Επίτροπε, θα ξεκινήσει λοιπόν η Επίτροπος. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε μια ακόμα ανταλλαγή απόψεων για το θέμα της ε, ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής Ευρωπαϊκής Ένωσης είπα. Πρόκειται για ένα νέο πλαίσιο προστασίας για την μεταφορά δεδομένων για εμπορικούς σκοπούς. Πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό και πολύ πιο ισχυρό πλαίσιο σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο του Safe Harbor, ε, το οποίο ακύρωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το περασμένο φθινόπερο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε ε, προσεκτικά την ασπίδα προστασίας και είμαστε πεπισμένοι ότι θα έχει υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένα. Την Παρασκευή τα κράτη-μέλη εξέφρασαν ε, συνολικά την ε, έγκρισή τους. Ε, το τελευταίο διάστημα εργαζόμαστε ακάματα με τις εταίρους μας από πλευράς ΗΠΑ για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις συστάσεις του Νοεμβρίου του 2013 και από τον περασμένο Οκτώβριο καθορίστηκαν και τα κριτήρια από το ε, δικαστήριο στην απόφασή του για το Safe Harbor. Η νέα σπίδα προστασίας συμμορφούνται προς αυτά τα κριτήρια και τις συστάσεις και ξεπερνά τις αδυναμίες της προηγούμενης συμφωνίας του Safe Harbor. Εγώ ε, σας απίθυνα το λόγο στις 13 ε, ε, Μαΐου, μία μέρα πριν την έγκριση του ψηφίσματος για την ασπίδα προστασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άκουσα πολύ προσεκτικά τις απόψεις σας και τις απόψεις που εξέφρασαν και άλλοι ενδιαφερόμενοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σας. Το ψήφισμα μαζί με τη γνωμοδότηση των αρχών ε, ε, προστασίας δεδομένων στην ομάδα εργασίας 21 οδήγησε σε σημαντικές διευκρινήσεις και ενίσχυσε περαιτέρω την ασπίδα προστασίας. Τι έχουμε καταφέρει. Καταρχάς, το θέμα της ε, ε, συλλογής δεδομένων. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι κεντρικό ε, θέμα συζήτησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταφέραμε να έχουμε κάποια επιπλέον αποτελέσματα. Έχουμε περαιτέρω εξασφαλίσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τους περιορισμούς και τις δικλείδες ασφαλείας κατά την εφαρμογή αυτή της μορφής. Καταρχάς, η συλλογή δεδομένων ε, θα χρησιμοποιείται ε, κατ' εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση μόνο όταν είναι στοχευμένη και δεν μπορούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο ύποπτο μόνο. Δεύτερον, θα εφαρμόζονται φίλτρα και άλλα εργαλεία ώστε να επικεντρωθούμε σε συγκεκριμένες ε, ανάγκες εθνικής ασφαλείας και να περιορίζουν τα δεδομένα που συλλέγονται και τρίτον, αυτό αφορά μόνο ένα κλάσμα της ε, μεταφοράς δεδομένων που γίνεται ε, μέσω διαδικτύου. Αυτές ε, οι διασφαλίσεις επιτρέπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι δραστηριότητες των υπηρεσιών εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι στα πλαίσια αυτών των οποίων θεωρούνται ως απαραίτητες και αναλυγικές λύσεις. Είναι ο έλεγχος ο οποίος θα πρέπει να γίνεται όταν προσπαθούμε να έχουμε αντίστοιχο επίπεδο προστασίας με βάση και το κατώτατο όριο που έχει θέσει το δικαστήριο. Αυτό όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων. Τώρα, ο μηχανισμό ε, του Ombudsman. Εδώ έχουμε περαιτέρω διασφαλίσει ότι θα ενισχυθούν και θα διευκρινιστούν τα βασικά σημεία που ανησυχούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλου ενδιαφερομένου. Εδώ να σας ε, το επισημάνω ότι και οι συζητήσεις που κάνατε ε, με σημαντικούς εταίρους στην Washington επέτρεψαν να προχωρήσουν τα πράγματα περαιτέρω και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό σήμερα. Τι καταφέραμε εδώ. Καταρχάς έχουμε περαιτέρω διασφαλίσεις για την ε, λειτουργική ανεξαρτησία του ε, Ombudsman. Επίσης υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις ότι πέραν της πλήρης ανεξαρτησίας του από την υπηρεσία ασφαλείας, ο Ombudsman θα διεξάγει τα καθήκοντά του ε, χωρίς καμία επιρροή η οποία θα μπορούσε ίσως να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της ανάλυσης του. Επίσης, διευκρινίσαμε τον τρόπο με τον οποίο ο Ombudsman θα συνεργαζεται με άλλους ανεξάρτητους ε, ε μηχανισμούς εποπτείας ε, των ΗΠΑ που έχουν συγκεκριμένες εξουσίες ε, και έχουμε διευκρινίσει ότι θα λαμβάνονται μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες για να διεξάγει τα καθήκοντά του ο και για να μπορέσουμε να έχουμε και διευκρίνηση της κατάστασης. Όπως ξέρετε, στον τομέα της εθνικής ε, ε, ασφάλειας οι αποζημιώσεις ε, είναι περιορισμένες, όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και στα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θέλουμε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό που θα αντιμετωπίζει τις καταγγελίες για πρόσβαση σε θέματα εθνικής ασφαλείας. Αυτή επεκτείνεται και σε όλα τα προσωπικά δεδομένα και σε όλες τις μορφές ε, εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως και δεδομένα τα οποία μεταφέρονται από άλλα ε, εργαλεία όπω για παράδειγμα ρήτρε για συνεργασία με τρίτου. Αυτό θα προσδώσει και ασφάλεια δικαίου για όλε τι ε, διαβιβάσει δεδομένων προς τι ΗΠΑ. Ο Ombudsman είναι μια πολύ σημαντική καινοτομία. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης μεμονωμένων καταγγελιών στον τομέα αυτό σε διεθνές επίπεδο. Σας ε, προτρέπω λοιπόν να μην ε, ε, απορρίψετε αυτό το μηχανισμό πριν ελεγχθεί η εγκυρότητά του. Λάβετε υπόψη ότι υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία και πιθανά ωφέλη. Να τους δώσουμε μια ευκαιρία και από εκεί και πέρα να είμαστε υπόλογοι να αποδείξουμε ότι όντως στην πράξη έχει αποτελέσματα. Τρίτον, όσον αφορά το θέμα της διατήρησης των δεδομένων, τώρα υπάρχει πλέον ρητή υποχρέωση για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ να διαγράφουν τα προσωπικά δεδομένα, αυτή τη στιγμή δεν απαιτούνται πλέον για, τον, για το σκοπό της επεξεργασίας. Αυτό ανακλά αυτό που έχουμε στην παρούσα και στη μελλοντική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων μας. Τέταρτον, έχουμε ενισχύσει περαιτέρω τους κανόνες ε, για τις ε, διαβιβάσεις, ε, ώστε η ασπίδα προστασίας να μην μπορεί να παρακαμφθεί μέσω διαβίβασης ε, δεδομένων Ευρωπαίων σε άλλους, ε, είτε στις ΗΠΑ είτε οπουδήποτε αλλού. Πέμπτον, όσον αφορά τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνει καταγγελία ε, ένας ε, πολίτης μεμονωμένα, ε, εξηγήθηκε καλύτερα η δυνατότητα και βάσει της απόφασης διευκρινίζεται ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να εξαντληθούν όλες οι ε, διαδικασίες αυτές ώστε να μπορέσει να αποζημιωθεί κάποιος πολίτης. Επίσης να σας πω ότι στο παρελθόν πάνω από το 90% αυτών των καταγγελιών για προστασία δεδομένων όπως ε, αιτήματα για διαγραφή ή για διόρθωση αντιμετωπίστηκαν με απευθεία επαφή με τις επιχειρήσεις. Και ελπίζουμε ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνεται τώρα, αλλά θα είναι ακόμα πιο εύκολο, διότι έχουμε ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ ε, των αρχών επιβολής ε, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, που σημαίνει ότι οι, προστασ... οι υπηρεσίες προστασίας δεδομένων και η Επιτροπή Εμπορίου και το Τμήμα Εμπορίου το αντίστοιχο τη ε, αμερικανική πλευρά. Ε, θα υπάρχει ένας οδηγός από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα εξηγεί αναλυτικά τα δικαιώματα που έχει ο καθένας βάσει της ασπίδας προστασίας. Επίσης, οι Ηνωμένε Πολιτείες πρέπει να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε εξέλιξη η οποία θα αμφισβητεί τη λειτουργία της ασπίδας προστασίας και αυτό φυσικά θα συνεισφέρει και στην ετήσια κοινή αναθεώρηση στην οποία θα συζητούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες τη λειτουργία του πλαισίου. Αυτή η κοινή αναθεώρηση ε, όπως θα θυμάστε, θα καλύπτει όλες τις πτυχές του πλαισίου και θέματα εθνικής ασφαλείας και μηχανισμούς αποζημιώσεων, όπως για παράδειγμα και το θέμα του Ombudsman. Θα ε, περιλαμβάνει και τη συμμετοχή των κατάλληλων φορέων, όχι μόνο από πλευράς ΗΠΑ, αλλά και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα τις αρχές προστασίας δεδομένων μας. Θα ε, αναφέρουμε τις διαπιστώσεις μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και από εκεί και πέρα μπορούμε να συζητήσουμε και ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είμαι ανοιχτή προς αυτό, θα μπορούσατε ίσως να ορίσετε κάποιον ο οποίος ε, θα είναι συνδεδεμένος με τα θέματα της κοινή αναθεώρησης της ασπίδας προστασίας. Τονίζω πάντα ότι μία από τις βασικές διαφορές μεταξύ της ασπίδας προστασίας και του safe harbor είναι ότι η ασπίδα προστασίας είναι μια δυναμική διαδικασία εν εξελίξη και εγώ δεσμεύομαι να παρακολουθώ τακτικά την ασπίδα προστασίας και θα διασφαλίσω ότι αυτό θα γίνεται και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η δέσμευση αυτή επίσης ε, ε, υποστηρίζεται και από μια πολύ αυστηρή ρήτρα αναστολής, την οποία θα χρησιμοποιήσουμε, να είστε βέβαιοι γι' αυτό, αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν ε, κενά από πλευρά ΗΠΑ και από πλευρά κυβέρνηση και από πλευρά επιχειρήσεων και δεν μπορούν να τηρήσουν τα υπεσχημένα. Ελπίζουμε λοιπόν να μην μείνει ξεχασμένη σε ένα σιρτάρι Έχουμε καθήκον και ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι μια τρίτη χώρα θα συνεχίσει να σέβεται τις υποχρεώσεις της, θα παρέχει αντίστοιχο επίπεδο προστασίας στα προσωπικά μας δεδομένα, όπως εμείς διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα των δικών τους πολιτών ε, προστατεύονται πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ασπίδα προστασίας ε, προσφέρει ε, πλήρη προστασία και πολύ ισχυρή ευθύνη. Επίσης, η απόφαση διευκρινίζει ότι θα αξιολογήσουμε το επίπεδο προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας μετά την έναρξη εφαρμογής ε, του κανονισμού για τη γενικότερη προστασία δεδομένων. Συνοψίζοντας, ε, η αναθεωρημένη ασπίδα προστασία τη ιδιωτική ζωή Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυστηρότερου κανόνε για τι αμερικανικέ επιχειρήσει για τη χρήση και ε, επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνουν. Επίσης, ενεργός εφαρμογή από τις Αμερικανικές Αρχές, συγκεκριμένες δυνατότητες ε, αποζημίωσης ε, και ε, ανάκλησης για συγκεκριμένους πολίτες και τέταρτον διασφάλιση για τις περιορισμούς και τις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζονται για τη χρήση προσωπικών δεδομένων για λόγους προσωπικής ασφαλείας και ε, στους σκοπούς επιβολής του νόμου. Και πέμπτον, τακτικές κοινέ αναθεωρήσεις με ε, συνεχή παρακολούθηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ασπίδα προστασίας λοιπόν έχει ενισχυθεί περαιτέρω όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, την ομάδα εργασίας του άρθρου 39 συνάδει πλέον με την απόφαση FREMS και υπάρχει πλήρης υποστήριξη από πλευράς κρατών μελών. Βάσει της αξιολόγησής μας, η ασπίδα προστασίας διασφαλίζει ισότιμο επίπεδο προστασίας και ελπίζω ότι όταν διαβάζετε τα έγγραφα της ασπίδας προστασίας θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πιστεύω ότι πλέον πρέπει να λάβουμε μια απόφαση και από εκεί και πέρα η ασπίδα προστασίας θα πρέπει να δοκιμαστεί επειδή υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ασπίδα προστασίας για την ε, ευρωπαϊκή οικονομία και για τις επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους καταναλωτές που βασίζονται ως στη δυνατότητα να μεταβιβάζονται δεδομένα προς τις ΗΠΑ. Θα καλύψει το νομικό κενό το οποίο υπάρχει μετά από την ακύρωση του Safe Harbor ε, πριν από 7 μήνες και θα υπάρχει προστασία και ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις. Εσείς, ε, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαδραματίσατε πολύ σημαντικό ρόλο ε, στη συζήτηση που έγινε τα τελευταία χρόνια για τις ε, μεταφορές δεδομένων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γι' αυτό. Σας ζητώ να συνεργαστείτε μαζί μου προκειμένου να είναι υπετυχημένο αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Um, ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε τους συναδέλφους με τη σειρά που ζήτησαν το λόγο. Παρακαλώ κανένα δίλεπτο ο καθένας. Κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω ότι για την Επιτροπή όλα αυτά είναι σημαντικό να έρθουν στο προσκήνιο και να συζητηθούν πριν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάποια πράγματα πρέπει να βελτιωθούν, ιδιαίτερα όσον αφορά τη συλλογή κάποιων δεδομένων με τρόπο συλλογικό το θέμα του Ombudsman ή της Ombudsfrau, όπως λέει στα γερμανικά, της γυναίκας δηλαδή διαμοσλαβητής, το θέμα επίσης της ασπίδας και των διαφορών μεταξύ του Safe Harbor και της προστασίας. Το Working Party 29. Από τον Απρίλιο μέχρι τώρα έχει συζητηθεί και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το κομμάτι το εμπορικό και το οικονομικό. Ξέρω όμως ότι μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει τίποτα, μπορεί να μας πει η Επίτροπος αν ξέρει κάτι καινούριο. Επίσης η οδηγία του 95 είναι αυτή που έχει ουσιαστικά αποτελέσει τη βάση για αυτήν την ασπίδα, για αυτήν την ε, προστασία. Θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται όμως με τα νέα δεδομένα. Υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία για το υπάρχον κείμενο. Ξέρω ότι κάποιοι δεν είναι πολύ ευτυχείς τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη έχουν ήδη κάνει κάποιες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων. Τις έχετε, μπορείτε να μας τις ε, δώσετε και μας. Ευχαριστώ που υπήρξατε σύντομοι. Ο κ. Βος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο, καταρχήν, που μας έκανε αυτή την παρουσίαση. Αν συγκρίνω αυτά που λέτε με τους στόχους μας, τους στόχους του ΕΛΚ, της πολιτικής μας ομάδας, εμείς θέλουμε βεβαίως ε, να εξαλειφθεί αυτός ο μηχανισμός Safe Harbor και γνωρίζουμε ότι αυτά που προτείνει και συμπεριλαμβάνει δεν αρκούν. Θέλουμε ελεύθερη ροή των πληροφοριών, με την σωστή παρακολούθηση και βεβαίως να κοιτάξουμε όλα τα θέματα που άπτονται του ανταγωνισμού, ιδιαίτερα σε εμπορικέ σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Σας ευχαριστώ γιατί μας παρουσιάσατε αυτούς τους στόχους με ικανοποιητικό τρόπο. Τίποτα βέβαια δεν είναι τέλειο. Υπάρχουν σίγουρα 2, 3, 5% στοιχείων που θα θέλαμε να συμπεριληφθούν που λείπουν, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό που προτείνεται σίγουρα είναι μια σημαντική βελτίωση του Safe Harbor. Επίσης θεωρώ ότι η ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας που θα πρέπει πάντα να εξετάζονται με ισορροπημένο τρόπο έγιναν βάσει της τελευταίας σας πρότασης προσεκτικά. Ξέρουμε επίσης ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζήτησε να υπάρχει προσεκτική προσέγγιση γνωρίζουμε και τις νομικές συνέπειες, γνωρίζουμε και ποια είναι τα μέσα που μπορεί να επικαλεστεί κανείς εάν υπάρχουν ανάγκες για προσφυγές, αν παραδείγματο χάρη η πρόσβαση σε δεδομένα δεν είναι μια πρόσβαση η οποία επιτρέπεται Ξέρουμε ότι οι δυνατότητες προσφυγής είναι ελάχιστες και θα ήθελα να σας συγχαρώ γιατί αυτό που προτείνετε είναι ίσως το πιο αποτελεσματικό που θα μπορούσαμε να προτείνουμε έναντι των πιθανών ε, αν θέλετε προτάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το Alternative Dispute Redress σε σύγκριση με το Privacy Shield Panel που υπάρχουν διαφορές. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι διαφορές για να κατανοήσουμε και εμείς καλύτερα ότι εμείς σαν Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε τέσσερα ή πέντε διαφορετικά επίπεδα προστασίας των δικαιωμάτων μας και των δεδομένων μας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ιντεβελτ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σίγουρα η πρόταση που έχουμε μπροστά μας, ή μάλλον η διευθέτηση αυτή, είναι καλύτερη από τις ασφαλείς λιμένες του Safe Harbor. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα Κατά πόσο αρκεί η πρόταση είναι το ζήτημα. Όπως και ο πελελής σα εξεπλάγει από την αξιολόγηση του κ. Φως που είναι νομικός. Δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ νόμου και εμπορικών συμφερόντων. Πρέπει να συμμορφώνεται κανεί με τον νόμο. Τελεία και παύλα. Αν δεν σα αρέσει ο νόμο, πρέπει να αλλάξει τον νόμο. Δεν εκφράζεται μια απλή πολιτική άποψη σε μπαρ είναι θέμα πολιτικής ε, δικαιοσύνης. Από το νότο δικαστήριο είναι αυτή, χρειάζεται αυτή η άποψη. Κύριε Επίτροπε, έχουμε αποκλίνουσε απόψει. Δεν είμαι νομικός. Δεν μπορώ να κρίνω. Αλλά δεν πείθομαι, δεν θεωρώ ότι αυτό εδώ αντιμετωπίζει τα προβλήματα που με το ΣΡΕΜΣ. Ο κ. ΣΡΕΜΣ και κάποιο άλλο, εγώ πιστεύω, θα προσφύγουν στο δικαστήριο. Και θα ξαναυπάρξουν προβλήματα. Θέλουμε ασφάλεια δικαίου που θα αντιμετωπίζουν και οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μας και δεν τους δίνουμε ασφάλεια δικαίου. Υπάρχει κάποια βεβαιότητα που πλανάται ε, και αυτό δυσχεραίνει την επιχειρηματικότητα. Ας διερωτηθούμε. Αν θεωρήσουμε ότι αυτό είναι το πρότυπο, είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε παρόμοιες λύσεις σε άλλους εμπορικούς εταίρους όπως η Κίνα και η Ρωσία. Εγώ δεν είμαι σίγουρη. Είμαστε πρόθυμοι να συναλλαγούμε μαζί τους υπό παρόμοιες συνθήκες. Πολλές ερωτήσεις ετέθησαν. Περιμένω απάντηση στην εξή ερώτηση. Ποιο είναι το νομικό καθεστώς των διαβεβαιώσεων που παρουσιάστηκαν. Είναι διακηρύξεις προεδρικές ε, ε, και κάθενας ε, δίνει κάποιες υποσχέσεις. Αν οι Αμερικανικές αρχές είναι σοβαρές και έχουν δεσμευτεί. Γιατί δεν θεσπίζουν μια νομοθεσία για να μας δώσουν ασφάλεια δικαίου. Υπάρχει δισταγμός και δεν δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνη. Άλλο θέμα εμπιστοσύνη για το συνήγορο του πολίτου. Έχουμε ένα πρότυπο. Μεταξύ αυτών ανεξάρτητη αρχή θέλουμε. Εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες φάει την εξαρτησία του διαμεσολαβητού. Διότι δεν την αποκαλούν διαμεσολαβητή, ανώτατο συντονιστή για, διεθνής, ε, για διεθνή διπλωματία για θέματα πληροφορικής. Διπλωματία. Μπορεί να προσφύγει κανείς εδώ και να διεκδικήσει δικαιώματα σαν πολίτης. Η κυρία Νοβέλη, η νέα ε, διαμεσολαβήτρια ή υπεύθυνη για διπλωματία δεν θέλει να έρθει να μας εξηγήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς βλέπει τα καθήκοντα πρέπει να εκτελέσει. Θα ήταν πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο με τη διευκρίνηση για δημιουργία κλίματος ε, εμπιστοσύνη. Τώρα για τη μαζική συλλογή δεδομένων. Αυτό είναι το βασικό θέμα, η καρδιά του θέματος. Παρά τις διαβεβαιώσεις που έχουμε. θεσπίσαμε νέα νομοθεσία. Πρέπει να διερωτηθούμε. Θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προδιαγραφές αυτές ή δεν παίρνουμε τους εαυτούς μας σοβαρά. Τέλος, είπα το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την κοινή αποτίμηση. Καλή πρόθεση αυτή, αλλά δεν είναι καλή ιδέα. Θα δεσμευτούμε τι το τρόπος. Από ρήτρες Άρα ποτέ δεν θα μπορέσουμε να ασκήσουμε αποτελεσματικό έλεγχο. Από προσωπική εμπειρία, επειδή με 12 χρόνια ευρωβουλευτή έχουμε ποτέ ασκήσει σοβαρά κάποια κριτική όσον αφορά τις αποτιμήσεις για τη συμφωνία SWIFT, για το PNR και όλα τα άλλα θέματα που πρέπει να ελέγχουμε. Ποτέ δεν ασκούμε σοβαρό έλεγχο. θα πρέπει να ελέγχουμε την αποτίμηση αυτή την αναθεώρηση και όχι να συμμετάσχουμε. Καταλαβαίνω τον πειρασμό, συνάδελφοι, να αναφερθείτε στις λεπτομέρειες, αλλά έχουμε στις 17 και 30 την κοινή συζήτηση Έκον Λίμπε. Παρακαλώ να είστε λακωνικοί. Γιάννα Ολμπρέχτ. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρουσίασή σας, για την εργασία που έχει κάνει η Επιτροπή μετά την ακύρωση από μέρους του δικαστηρίου της απόφασης για το Safe Harbor. Εμείς από την αρχή μιλήσαμε για αυτό το καθεστώς παρανομίας τα τελευταία 15 χρόνια και καταρχήν θα πρέπει να πούμε ότι βεβαίως θα πρέπει να επανέλθει η εμπιστοσύνη των πολιτών όσον αφορά το νόμιμο και ασφαλές σύστημα προστασίας. Πρέπει να μας εμπιστεύονται και να έχουν και εμπιστοσύνη στην προστασία που ενδεχομένως μπορεί να τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα δεν είναι οι βελτιώσεις. Το θέμα είναι αν εδώ συμμορφωνόμαστε με το κοινοτικό δίκαιο, όπως καθορίζεται από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης, η τελευταία απόφαση και δεν θα επανέλθω επαναλαμβάνοντας αυτά που είπαν προηγούμενοι ομιλητές, αλλά όσον αφορά αυτή την ε, μαζική συλλογή δεδομένων, Αυτό θα πρέπει να αποκλειστεί από αυτήν την απόφαση. Η κάθε πληροφορία δεν μπορεί να συλλέγεται. Γιατί βεβαίως εδώ βλέπουμε ότι λιγότερα δεδομένα συλλέγονται από μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει, ναι, δεν τα συλλέγουμε όλα, όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στον κόσμο. Ναι, απ' την άλλη όμως ε, αυτά που συλλέγονται είναι ήδη αρκετά, ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι από τη μία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διαπιστώνει στην αποφασή του ότι δεν αρκεί εδώ το, ε, η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τίποτα δεν αλλάζει έτσι και αλλιώ στην νομοθεσία των ΗΠΑ και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα έτσι και αλλιώς να αλλάξει. Άρα, εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε αυτές οι βελτιώσεις που προτείνονται εδώ αν αρκούν. Όμως, ο έλεγχος δεν σημαίνει ότι θα αρχίσει να ισχύει για πάντα αυτή η νομοθεσία. Ας πούμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι θα το δοκιμάσουμε, θα το ελέγξουμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Αν δεν αρκεί αυτή η προστασία, θα πρέπει να επανέλθουμε στη διαπραγμάτευση και να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Έτσι κι αλλιώς για τον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει κανένας κανόνας για την προστασία των δεδομένων στις Ηνωμένε Πολιτείες. Στις όπου θα μπορούσε να εφαρμοστεί το Safe Harbor, έτσι και αλλιώ σε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν θα εφαρμοστεί. Στις Ηνωμένε Πολιτείε υπάρχουν ομάδε της κοινωνίας των πολιτών που επιθυμούν, όπως και εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να βελτιώσουν τα πράγματα. Αφού λοιπόν και εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε τα πρότυπα που θα διέπουν τις ε, σχέσεις μας με τις Ηνωμένε Πολιτείε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να συμπεριλάβουμε και εκεί κάποιες τέτοιες προτάσεις. Αλλιώς θα υπάρξει νέα απόφαση του δικαστηρίου καταδικαστική και πάλι θα χάσουμε εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Πρόεδρος. Κοιτάξτε, εμείς είχαμε καλέσει την κυρία Νοβέλη, αλλά όχι επίσημα. Πρέπει να είμαστε δίκοι λοιπόν. Ωραία, γιατί δεν το κάνουμε, γιατί δεν την καλούμε επίσημα. Θα το υποβάλλω στους συντονιστές. Κύριε Άλμπρεχτ, έχετε διαδικαστικό. Όχι. Κύρκο, ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε. Έτσι και αλλιώς υπάρχουν πολιτικές ομάδες που σε καμία περίπτωση δεν θα ικανοποιηθούν με καμία συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτης χώρας. Και εγώ είμαι νομικός και όσον αφορά την νομική σας εξήγηση την θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα. Πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το πιο θετικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι αποφάσεις, αυτό το νομικό πλαίσιο, παραδείγματος χάρη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι το 60% αυτών που αφορά η απόφαση αυτή, αλλά και το safe harbor. Θα πρέπει λοιπόν όσον αφορά αυτόν τον συνήγορο του πολίτη, αυτό τον ombudsman, η άντρας η γυναίκα πρόκειται, ο συγκεκριμένο ρόλος του νομίζω ότι θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά. Δεν είμαι διατεθειμένος εγώ να το εγκαταλείψω αυτό το θέμα χωρί να το συζητήσουμε. Επίσης, το θέμα των... Ε, όσον αφορά τα δικαιώματα αποζημιώση κάλυψη, τα redress rights και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί στο γενικότερο πλαίσιο των σχέσεών μας με τις ΗΠΑ το θέμα της ε, μαζικής ε, συλλογής δεδομένων. Εδώ σε κάθε περίπτωση οι Ηνωμένε Πολιτείε στέλνουν ε, αποφάσεις σαν πυράβλους κατά ημών και η σημασία τους αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντική. Όσον αφορά λοιπόν το διάταγμα αυτό για τις αποζημιώσεις. Έχουν υποβληθεί οι προτάσεις του Κοινοβουλίου και αυτή η πρόταση για την ασπίδα προστασία σίγουρα καλύπτουν τα κενά της προηγούμενης νομοθεσίας, αλλά δεν είναι δυνατόν εδώ να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την εμβέλεια των αποφάσεων και της νομοθεσίας των ΗΠΑ χωρίς να δείξουμε δικές μας προτάσεις. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε γιατί η εργασία σας είναι εξαιρετική σε πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Και η παρουσία σας εδώ σήμερα είναι εξαιρετικά χρήσιμη για μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να είμαι ειλικρινής. Κυρία Γιώροβα, είστε σήμερα εδώ και μας ενημερώνετε για το τελικό αποτέλεσμα, την τελική πρόταση. Βεβαίω θα μπορούσατε να το κάνει και λίγο πιο νωρί. Γιατί εμεί θα θέλαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είχε λίγο νωρίτερα τη δυνατότητα να εκφραστεί, να επεξεργαστεί. Εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία είναι ικανοποιητική και συζητήσαμε μέσω των συντονιστών με έντονο τρόπο το θέμα αυτής της διαδικασίας. Ξέρετε πολύ καλά ότι πρόκειται για ε, λεπτό θέμα για μας και θα πρέπει να το πάρετε σοβαρά. Θα ήθελα πολύ να μας παίρνατε λίγο πιο στα σοβαρά και να μην έρχεστε εδώ μόνο για να ανταλλάξουμε ευγενικά σχόλια. Για μένα είναι απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Αν θέλετε, δεν μου φαίνεται ότι πρόκειται για πραγματική επιτυχία. Εντάξει, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, αλλά στην πράξη δεν προστατευόμαστε. Και βεβαίως αρχές ε, ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών θέλουν να μας προστατεύσουν. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται με τον ε, Ombudsman, το πρόσωπο που θα αναλάβει αυτήν την θέση. Αν διαβάσω στο παράρτημα, μα δεν έχει νομικά μέσα. Τι μπορεί να κάνει. Όλη αυτή η ιδέα, αν θέλετε, αυτού του ατόμου είναι εξαιρετικά σαφής η ανεξαρτησία των αρχών επιτήρησης επίσης. Και αυτό συζητείται πολύ. Και το τελευταίο σημείο, το οποίο το είχαμε συζητήσει και τίποτα δεν άλεξε, είναι το θέμα της προστασίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση του κοινοτικού δικαίου. Δεν είναι δυνατόν να τους χωρίσουμε σε αυτούς οι οποίοι είναι Ευρωπαίοι πολίτες και δεν είναι παραδείγματος χάνει κάποιος περνάει τις διακοπές του, τις καλοκαιρινές. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμμορφωθεί και δεν συμβαδίζει με το κοινωτικό δίκαιο. Και διαβάστε προσεκτικά την απόφαση του δικαστηρίου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπόν και η κυρία Γκόμη είπαν ότι δεν θα μιλήσουν για να μας βοηθήσουν. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Ο κύριος Λόπεθ Αγγιλάρ. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Οι δικέ μου ανησυχίε συνάδουν με κάποια από τα πράγματα που ακούστηκαν. Αυτό όμως το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι αφού παραδεχτούμε ότι υπάρχει κάποια πρόοδος σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία του Safe Harbor. Καταρχάς, πόσα από αυτά θα εξαρτηθούν από την αποτελεσματικότητα των προεδρικών διαταγμάτων, τα οποία γίνονται για να διασφαλίσουν ότι θα εφαρμοστεί αυτό το νέο πρόγραμμα, δεδομένου ότι έχουμε και επερχόμενες προεδρικές εκλογές και μπορούν να ανατραπούν τα πάντα από αμερικανικής πλευράς. Αν δεν υπάρχει δεσμευτική νομοθεσία η οποία θα εφαρμόζεται και από τις δύο βουλέ του Κογκρέσου. Τα πάντα θα εξαρτώνται από τη βούληση του Προέδρου ε, για να ε, συνεχίσει να ισχύει. Και δεύτερον, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι να διασφαλίσουμε ότι θα δίνεται ερμηνεία ε, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας βάσει της Χάρτας των Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων. Αλλά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλάζει. Η διαδικασία είναι δυναμική διότι υπάρχει μια νέα δεσμή μέτρων για την προστασία δεδομένων η οποία θα τεθεί σε ισχύ και πόσο από αυτά θα συμπεριληφθούν ε, για να εξυπηρετήσουν και την αποτελεσματικότητα του νέου προγράμματος. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ, συνάδελφοι, για την υπομονή σας, ε, δεδομένου ότι είχαμε πολύ λίγο χρόνο στην ε, διάθεσή μας. Κύριε Επίτροπε, αυτές είναι οι ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Θα ξεκινήσω με τις ερωτήσεις της κυρίας Σίπελ. δεχτήκαμε τις συστάσεις της ε, ομάδας εργασίας του άρθρου 29 και προς έκπληξή μου ήταν πολύ πιο δύσκολο από τις συστάσεις για την εθνική ασφάλεια. Αυτή βέβαια είναι η εντύπωση που έχω εγώ για αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων. Δεχτήκαμε λοιπόν τις συστάσεις για τη διατήρηση των δεδομένων, ε, για τις ε, ε, μαζικές ε, ε, διαβιβάσεις. Ζητήσαμε να περιληφθούν και οι χώρες ΟΧ, Λίχτενστάιν, Ισλανδία και έχουμε συμπεριλάβει και την αυτόματη λήψη αποφάσεων. Συμπεριλαμβάνεται και αυτό στις συστάσεις των αρχών προστασίας δεδομένων και επίσης να αλλάξουμε τις δυνατότητες προσφυγής για τους πολίτες. Θεωρώ λοιπόν ότι αντιμετωπίσαμε και ασχοληθήκαμε με όλες τις βασικές συστάσεις και τα έχουμε όλα πλέον στο κείμενο της απόφασης. Η απόφαση και τα σχετικά έγγραφα έχουν υποβληθεί με βάση την οδηγία ενισχύ. Και συγγνώμη τώρα που μιλάω λίγο νομικιστικά, αλλά προσπαθήσαμε να έχουμε ισότιμη προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων πολιτών με βάση το παρόν ε, εφαρμοστέο δίκαιο, δηλαδή την οδηγία. Και βεβαίως έχετε δίκιο, δεν μπορούμε να ξεχνούμε ότι η ημερομηνία εφαρμογής του νέου κανονισμού είναι η 25η Μαΐου του 2018. Επομένως είναι πρώτον πυλών. Κάποιοι από εσάς το είπατε και ο κύριος Άλμπρεχτ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Πρέπει λοιπόν να γίνουν όλα σωστά. Διότι αυτή τη στιγμή η απόφαση αφορά την αυξημένη ζήτηση σε σχέση με την οδηγία κυρίως ε, τη διατήρηση των δεδομένων και τις ε, μαζικές ε, διαβιβάσεις και κάποια άλλα στοιχεία, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι. Θα πρέπει να είμαστε αυθεντικοί και να επιδείξουμε ισχύ και να συνεχίσουμε να πιέζουμε την αμερικανική πλευρά και ήδη ανακοινώσαμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κανονισμός για την προστασία των δεδομένων αποτελεί επανάσταση στην προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Αμερικανοί εταίροι μας το γνωρίζουν αυτό. Και θα ήθελα να τα δούμε από την πολύ πρακτική σκοπιά τα πράγματα. Εμείς θα δούμε τι γίνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές ε, για τον κανονισμό για την προστασία δεδομένων για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Συνεργαστήκαμε στενά με τις αρχές προστασίας δεδομένων που είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι αυτοί οι οποίοι αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει στην προστασία δεδομένων, πού έγκυνται οι κίνδυνοι και οι απειλές και θα συνεργαστούμε μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κοινή αναθεώρησης. Η μία θα είναι για το καλοκαίρι του 2017 και η άλλη για το καλοκαίρι του 2018 και θα συνεργαστούμε επίσης για την ασπίδα προστασίας υπό την έννοια των πιθανών βελτιώσεων ή τροποποίησεων. Αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αναφερόμαστε στην ασπίδα προστασίας, στην ανάγκη ασφάλειας δικαίου για τις επιχειρήσεις και στην ομοθεσία όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, όταν γίνονται αλλαγές οι οποίες έχουν καλές προθέσεις, ε, παραδεχόμαστε κάτι αρνητικό στην πραγματικότητα. Επομένως, πρέπει να ε, φροντίσουμε να διατηρηθεί με μια ασφάλεια δικαίου και ταυτόχρονα να εξετάσουμε και τι δυνατότητες έχουμε για να βελτιώσουμε το σύστημα προστασίας βάσει της ασπίδας προστασίας, ώστε να σχετίζεται και με το γενικότερο κανονισμό για την προστασία δεδομένων. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή. Αυτή βέβαια είναι η άποψή μου ως νομικός. Αν καθήκον μας είναι να έχουμε αντίστοιχη προστασία προσωπικών δεδομένων στις Ηνωμένε Πολιτείες με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, όταν θα τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός, ούτω ή άλλω θα πρέπει να το εξετάσουμε αυτό, γιατί θα υπάρχουν οι κανόνε στην Ευρώπη. Αυτό θα είναι λοιπόν το βασικό ε, καθήκον που σας αναλογεί μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης αναθεώρησης του 2017 και 2018. Σας υπόσχομαι ότι δεν θα εθελετηθούμε και δεν θα αφήσουμε τα πράγματα να συνεχίζονται και να διαιωνίζονται. Υπάρχουν έξι που απέχουν και υπήρχαν και σχόλια από τη Γαλλία και τη Γερμανία που λένε το εξή στην ουσία. Δεχόμαστε την παρούσα εκδοχή Έχουμε κάποιες ανησυχίες για το κατά πόσον είναι η βέλτιστη δυνατή ή αν υπάρχουν κάποια περιθώρια βελτίωσης. Ας τις δώσουμε μια ευκαιρία και ας την εξετάσουμε και να δούμε κατά πόσο μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, ποιες είναι οι λειτουργικές πλευρές και πόσο επιτυχή θα είναι η εφαρμογή της. Περισσότερο λοιπόν ε, μας ενδιαφέρει η πρώτη χρονιά λειτουργίας της ασπίδας προστασίας και θα ήθελαν σε ένα χρόνο να το επανεξετάσουν και να αξιολογήσουν το ζήτημα. Αλλά ούτως ή άλλως όλοι αυτό πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Βος ε, για την ε, παρατηρήσεις σας και τα καλά σας λόγια. Σίγουρα πρέπει να εξισορροπήσουμε τα συμφέροντα μεταξύ δύο πολύ σημαντικών προτεραιοτήτων, της ασφάλειας και της προσωπικής ζωής. Ε, και δεν θα πρέπει να το λησμονούμε αυτό. Και όσον αφορά τις επιχειρήσεις, για να απαντήσω και στη Σόφη Ινεντβελτ, η νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Αλλά δημιουργούμε επιπλέον αρμοδιότητες και καθήκοντα για τις επιχειρήσεις που απορρέουν από την νομοθεσία αλλά οι προϋποθέσεις και τα καθήκοντα και οι, οι αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που θα πρέπει να τηρήσουν οι επιχειρήσεις αποτελούν ένα επιπλέον επίπεδο. Επομένως πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου, θα πρέπει να δούμε και τις επιχειρήσεις, τι επιβάρυνση έχουν, τι είναι εφικτό, τι είναι αποδεκτό και το αναφέρετε και κάποιοι από εσά άλλωστε, αυτό δεν γίνεται κυρίως για τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις, για τις μεγάλους καρχαρίες της αγοράς, το κάνουμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο μέσο χωρίς ε, να ε, πληγούν από νέες προϋποθέσεις και υπερβολική επιβάρυνση. Μαζική συλλογή δεδομένων και τις άλλες δυνατότητες προσφυγής. Δεν ξέρω αν έχουμε άλλο χρόνο. Στην ουσία, έχουμε τη δυνατότητα καταγγελίας προς τις επιχειρήσεις που ε, βάσει στατιστικών στοιχείων είναι και στην πλειονότητά τους ε, ε, αυτό που, το οποίο γίνεται, το 96% επιλύεται σε αυτό το επίπεδο. Μετά υπάρχει δυνατότητα προσφυγή στο δικαστήριο. Εμεί θα του ζητήσουμε να ε, προσφεύγουν στην αρχή προστασία δεδομένων. Η πιο δύσκολη περίπτωση είναι όταν διαβιβάζονται δεδομένα προ τι ΗΠΑ και η καταγγελία γίνεται ε, στον εισαγωγέα των ΗΠΑ που δεν είναι στη δικαιοδοσία των αρχών προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ λοιπόν ο πολίτης μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, την υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου, της Federal Trade Committee και σε κάποια χρόνια θα υπάρχει ε, δυνατότητα διαιτησίας όπου έχουμε συμφωνήσει ότι θα υπάρχει και τεχνική υποστήριξη για τους Ευρωπαίους από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων, θα υπάρχει υποστήριξη από νομικούς και θα υπάρχει και η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ε, βίντεο διασκέψεις ε, με τη βοήθεια και πάλι των Αρχών Προστασίας Δεδομένων και ελπίζω ότι αυτό το πάνελ διαιτησίας θα είναι η ίστατη λύση και θα χρησιμοποιείται πάρα πολύ σπάνια. Τώρα, νομικό καθεστώς. Φυσικά θα ήταν πολύ πιο εύκολο, καλύτερο να έχουμε νομοθεσία. Το παραδέχομαι. Έχουμε τις επιστολές όπου τα θεσμικά όργανα, όχι οι συγκεκριμένοι πολίτες, ε, υπογράφουν τις επιστολές. Δεν υπογράφει κανείς με την προσωπική του ιδιότητα, αλλά υπογράφουν εκ μέρους της Αμερικανικής Διοίκησης. Επομένως, ε, τα όργανα δεσμεύονται να κάνουν αρκετά ώστε η ασπίδα προστασίας να παραμείνει για να προστατεύονται οι πολίτες και τα δεδομένα τους. Ακόμα και αν γίνουν οι εκλογές, οι εκλογές πάντα είναι μια στιγμή αβεβαιότητας. Δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Αλλά τέλο πάντων να ε, μείνω στα της των ΗΠΑ. Σαφώς και οι εκλογές ε, θα δημιουργήσουν ε, αβεβαιότητα, αλλά περιμένουμε να διατηρηθεί η συνέχεια από τις Αμερικανικές αρχές οι οποίες δεσμεύθηκαν μέσω επιστολών που υπογράφονται από τους πλέον υψηλά ιστάμενους. Άκουσα και πολλές ερωτήσεις για τον Ombudsman, το διαμεσολαβητή. Καταφέραμε να διευκρινίσουμε περαιτέρω τις αρμοδιότητες και εξασφάλιση για την ανεξαρτησία ε, του Ombudsman. Ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να απαντά στις καταγγελίες. Δεν θα υπάρχει καμία καταγγελία η οποία δεν θα την χάνει επεξεργασίας. Θα υπάρχει δικαίωμα να ε, ε, ανακρίνει τους γενικούς επιθεωρητές και να χρησιμοποιήσουν και άλλους διάλογους για να βρουν πληροφορίες και από εκεί και πέρα θα πρέπει να απαντούν στο άτομο το οποίο έχει υποβάλει την καταγγελία. Κατά πόσον υπήρχε συμμόρφωση ή μη συμμόρφωση. Επίσης, θα ε, εξηγεί κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και τι προτείνεται ως λύση. Επιπλέον θα έχουμε και ένα θέμα το οποίο θα εξεταστεί εκεί στην ετήσια αναθεώρηση και θα δούμε, θα έχουμε μια εικόνα για το κατά πόσον υπάρχουν προβλήματα με το θεσμό του διαμεσολαβητή. Αυτό είναι ένα νέο μέσο το οποίο παρέχεται ακριβώ για αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχουμε κάτι αντίστοιχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και εγώ θα επακρυπνώ για να δω πώς θα λειτουργήσει αυτό ο νέος ε, ρόλος ε, του Ombudsman. Α δείξουμε εμπιστοσύνη στην αρχή και να δούμε από εκεί και πέρα πόσο ικανοποιητική θα είναι αυτή η λύση εν τέλει. την κυρία Ένστ. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος στη διαδικασία. Ενημερώσαμε το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ε, πολιτικών ελευθεριών. Ε, δύο μέρες καθυστέρηση νομίζω ότι υπάρχει. Συγγνώμη αν υπήρχαν δύο ή τέσσερις μέρες καθυστέρηση, αλλά σας διαβεβαιώ ότι εγώ λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη μου το Κοινοβούλιο, όχι μόνο την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, αλλά και τις άλλες τρεις αρμόδιες επιτροπές στις οποίες πηγαίνω και εξηγώ τι ακριβώς κάνουμε. Δεν είμαι ικανοποιημένη, δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένη, ούτε χαρούμενη. Εγώ όμως ακολουθώ τη διαδικασία, αναλαμβάνω την ευθύνη, υπέγραψα την απόφαση ε, περί καταλληλότητας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τηρήσω όλες τις υποσχέσεις που σας έχω δώσει ε, και σε εσά και σε πολλούς άλλους ε, φορείς, που θα ελέγχουμε την εφαρμογή της ασπίδας προστασίας και αν δεν είναι αποτελεσματική, αν κάποιος ε, δεν τηρήσει αυτά τα οποία δεσμεύθηκε ότι θα τηρήσει, ε, θα ανασταλεί το σύστημα. Αλλά πιστεύω ότι θα έχει αποτέλεσμα, θα παρακολουθήσουμε και τις αλλαγές στην Αμερικανική νομοθεσία. Είναι και ένα από τα ερωτηματικά μας άλλωστε αυτό. Υπάρχει η ε, οδηγία για την ε, ε, προεδρική πολιτική το υπαριθμό 28 και ένα νέο νομοσχέδιο και θα θέλουμε να υπάρχει εύρος στην νομοθεσία στις ΗΠΑ στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Όπως είπα συνάδελφε θα έχουμε των συντονιστών της ΛΥΜΠΕ μετά από αυτή τη συνεδρίαση. Ακριβώς με αυτό το θέμα θα Σχοληθούμε, Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους της Επιτροπής ΕΚΟΝ που θα αρχίσουμε καθυστερημένα τη συζήτηση στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Παρακαλώ τους συναδέλφους να έρθουν εδώ συμπεριλαμβανομένου του κύριου Φέρμπερ, τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ.